So, liebe σας και πάλι συνάδελφοι. Μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση σήμερα το πρωί με τι πολλέ ψηφοφορίε, τώρα το απόγευμα θα περάσουμε σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων και στο σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη έχουμε τον οδικό χάρτη για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών ε, σε άνθρακα, ανθρακούχων εκπομπών. Το σενάριο για την προστασία του κλίματος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χαμηλών εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα βιομηχανία. Αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ώστε να συζητηθεί και η θέση του Ευρωκοινοβουλίου και να καθοριστεί η τοποθέτηση <clears throat> του Κοινοβουλίου. Έχουμε ένα εισηγητή, τον Chris Davis. Ο Chris Davis παρουσίασε ένα έγγραφο εργασίας για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Κύριε Ντέιβις, έχετε τον λόγο. Chris Davis, παρακαλώ. Thank you, Chairman, for... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και που μας δίνετε την ευκαιρία να το συζητούμε. Δεν έχουμε πολλούς συναδέλφους παρόντες, μεν, αλλά η ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο με το νέο ανέτος θα είναι ίσως η πιο σημαντική που θα έχουμε να ε, διεξεγάγουμε στο Κοινοβούλιο. Ο χάρτης πορείας λοιπόν, με χαμηλά επίπεδα ανθρακού εκπομπών, ε, θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, καλύψει κατά 80% του στόχους της για τις εκπομπές μέχρι το 2050 και μια μείωση έως το 2030 κατά 40%, 60% έως το 2040 είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις εκθέσεις που έχει εκπονήσει το Κοινοβούλιο ή έχει εξετάσει το Συμβούλιο και που ε, καταγράφεται τα όσα έχουν υποθεί για, το, για, τις, για τις ε, εκπομπές και τη μείωση κατά 80% το 2050 μέχρι το 2050. Παρόλα αυτά λοιπόν που λέγονται, ο μόνος στόχος που έχουμε απτώσει είναι μείωση κατά 20% στο 2020 από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, εάν υιοθετηθεί αυτός ο οδικός χάρτης και εγκριθεί, θα δώσει πορεία για νέους στόχους που θα πρέπει να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα αλλάξουν ολόκληρα στην την προσέγγιση στην υπόθεση αυτή. Τώρα, θα έλεγα πρόεδρε ότι το συγκεκριμένο αυτό έγγραφο έχει εντό εισαγωγικών παντγώσει σε επίπεδο συμβουλίου, βρίσκεται σε ένα διέξοδο δηλαδή. Ε, ό,τι και να πει το κοινοβούλιο δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλη πολιτική συνέπεια ή απήχηση γιατί μόνο με την έγκριση του συμβουλίου μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Όμω, εάν η εν λόγω έκθεση απορριφθεί από το κοινοβούλιο, και ύστερα από τη δράση που είχαμε αναλάβει και την πρωτοβουλία του, με την έκθεση του κυρίου Έκχαουτ τον Ιούνιο, εάν πει το κοινοβούλιο ότι δεν δέχεται να ακολουθεί στον δρόμο αυτό, τότε νομίζω ότι θα δείχναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει νόημα να κατατίθενται προτάσεις ε, και πρωτοβουλίες νέε εάν ε, το Συμβούλιο της παγώνει και το Κοινοβούλιο της απορρίπτει. Αυτό νομίζω θα οδηγούσε μια συλλήβδινη αλλαγή στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε να θέσουμε ερωτήματα προφανή που όμως νομίζω αποτελούν και το υπόβαθρο πολλών από τι αποφάσει που λαμβάνουν τόσο οι ευρωβουλευτέ όσο και οι υπουργοί. Το πρώτο εξ αυτών είναι το εάν πράγματι πιστεύουμε πως οι περισσότεροι ε, επιστήμονες ανά τον κόσμο έχουν δίκιο όταν λένε ότι η αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη που έχει προξενήσει ο άνθρωπο λόγω των ανθρωπινών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται, και, πραγματοποιείται ε, με ταχύτητα τους ρυθμούς όπως λένε. Αν συμβαίνει αυτό και αν το πιστεύουμε θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερως γιατί αυξήθηκαν πέρσι το 2010 κατά, κατά 16% οι εκπομπές ανά τον κόσμο, τεράστια ανάπτυξη χωρίς προηγούμενο και αν θυμάστε το πάνελ για τις κλιματικές αλλαγές πριν από μερικά χρόνια που έλεγε ότι θα πρέπει να ε, όχι να ε, μην επιτρέψουμε την αύξηση των εκπομπών, αλλά να συγκρατήσουμε αυτή την αύξηση έως το 2015. Προφανώς δεν πρόκειται να επιτύχουμε το στόχο αυτόν, με δεδομένο ότι παρουσιάζεται ακόμη αύξηση. Και αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά περισσότερο από 10% είναι αρκετά πιθανή. Εάν συνεχίσουμε στη πορεία αυτή ως εκ τούτου, δεν φαίνεται πουθενά ορατό το πέρας αυτών των αύξησεων εκπομπών. Βέβαια, ούτε όλοι οι ευρωβουλευτέ, ούτε όλοι οι υπουργοί, ούτε και όλοι βέβαια οι ψηφοφόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν με αυτή την θέση, ότι έχουν δίκιο δηλαδή οι ε, επιστήμονε. Και χαίρομαι που με τον κύριο Κράμερ, τον συνάδελφο εδώ, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει και να διαδώσουμε βέβαια τι ιδέε που συζητήσαμε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδραμείου σε όλου του συναδέλφου τη Επιτροπή μα, γιατί νομίζω ότι αυτό ε, αυτή η αμφισβήτηση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεύτερο ερώτημα. Εάν δεν υπήρχε διεθνή συμφωνία, εάν δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, συνεχίζουμε και μόνοι μας έστω. Αυτό που θα έλεγε ίσως, ε, θα, θα ονομάζαμε ίσως δίλημα της Πολωνίας, δηλαδή αυτό που θα μπορούσε η Πολωνία να ερωτήσει ε, ενώπιον της υποχρέωσης να κλείσει τις ε, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού από ε, άνθρακα, όταν η Κίνα την ε, κάθε ημέρα που περνάει ανοίγει νέες μονάδες παραγωγής άνθρακα την, για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με ραγδαίους ρυθμούς και αυτό ισχύει και για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία. Είναι ευστα... ευσταθές λοιπόν αυτό το δίλημα. Ταυτόχρονα όμως ε, η Κίνα έρχεται ε, ως πρωταγωνιστής και της πράσινης τεχνολογίας, της ανανεώσιμης τεχνολογίας. Μέσα σε αυτή τη νέα τεχνολογία λοιπόν εγγράφεται η παραγωγή των νέων ε, μονάδων παραγωγής από άνθρακα. Αλλά ξέροντας ότι δεν μπορεί το μέλλον μας βεβαίως να στηρίζεται στον άνθρακα, στην καύση του άνθρακα, Χρειάζομαστε ασφαλώς τεχνολογίες με χαμηλή περιεπτικότητα άνθρακα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει για να μην πω χάσει το παιχνίδι σε σχέση με, τις, με την ηλιακή τεχνολογία και την ηλιακή ενέργεια. Και ως εκ τούτου πρέπει εξάπατος να μην χάσουμε άλλο χρόνο, να μην χάσουμε άλλο το παιχνίδι. Το 60% λοιπόν των εκπομπών προέρχονται από την απελευθέρωση ατμόσφαιρα και την ε, καύση ε, αερίου και άνθρακα και έτσι πρέπει σε αυτό το σημείο να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ε, Εμεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν δίνουμε σαφή μηνύματα. Η Giro Electric, η οποία εκπροσωπεί τους περισσότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ετοιμάσει το δικό της οδικό χάρτη για τον άνθρακα, με προτάσεις αντίστοιχες με αυτές που βλέπουμε από την IPCC των ΗΠΑ και με δεδομένο ότι οι παραγωγοί ήδη έχουν ε, ετοιμάσει έναν οδικό χάρτη, νομίζω ότι είναι σαφές πως βλέπουν ρεαλιστικά δυνατότητες, ρεαλιστικές δυνατότητες για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αυτό μας λένε όμως είναι ότι χρειάζονται τα εξής δύο. Πρώτον πρέπει οτιδήποτε εργαλεία έχουμε στη θέση μας να τα αξιοποιούμε, να μην περιορίζουμε δηλαδή του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ως προς τη χρήση της πυρηνική ενέργειας ή ω προς την σύλληψη και αποθήκευση άνθρακα τεχνολογία αυτή όπου είναι δυνατόν γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει ανάγκη τέτοιων τεχνολογιών όπως στην Αυστρία που έχει μεγάλη εξάρτηση από τι ανανεώσιμε, ενώ άλλε χώρε μπορεί να τι χρειάζονται άρα δεν πρέπει να δέσουμε τα χέρια της ε, ε, βιομηχανία, τη παραγωγή δηλαδή ηλεκτρικού. Και δεύτερον, αυτό που μα λέει η βιομηχανία είναι ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματο ανταλλαγών ε, εκπομπών. Στόχος αυτού του συστήματος αρχικά ήταν να πέφτει κατά 1,4% η εκπομπή ε, αερίων από τις ε, βιομηχανικές μονάδες που εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα, κατά κύριο λόγο, αλλά και δευτερογενώς γενικότερα η μείωση <clears throat> της χρήσης της τεχνολογίας του άνθρακα, πράγμα όμως το οποίο δεν εξασφαλίζεται γιατί είναι τόσο χαμηλές τιμέ του άνθρακα που δεν υπάρχουν τα σχετικά κίνητρα για την ε, παραγωγή, για τη βιομηχανία. Και ξέρουμε ότι όταν είχαμε συστήσει το ETS, ε το σύστημα ανταλλαγών δηλαδή πριν από 4-5 χρόνια, είχαμε ε, υπόψη, ε, περιμέναμε ότι <clears throat> το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε με τιμές άνθρακα κάπου στα 30 ευρώ στον τόνο, ενώ τώρα είναι στα 15 περίπου. Και ως εκ τούτου και ενώ δεν έχει προβλεφθεί η αύξηση των τιμών των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα δηλαδή μέχρι το 2020, δεν έχει υποδοτικότητα το σύστημα αυτό. Άρα δεν μπορούμε να... <clears throat> Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην πορεία αυτή. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές του άνθρακα <clears throat> του διοξιδίου καλύτερα του άνθρακα, του στόχου της μείωσης, να το, στόχο της μείωσης να τον περιορίσουμε ακόμη περισσότερο, δηλαδή να ξεπεράσει τον 1,4% και έτσι να υπάρξει το σχετικό κίνητρο, το αυτόματο κίνητρο για την ανάπτυξη τη επένδυση από πλευρά τη βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει αμέσω να ε, ενισχύσουμε του στόχου αυτού, να καταστήσουμε πιο αυστηρού του στόχου για να πιέσουμε τη βιομηχανία, αλλά ίσω θα έπρεπε τουλάχιστον στην τέταρτη περίοδο του ETS, το 2020-2025, ακόμα και το 2030, να έχουμε αυτού του στόχου κάποια στιγμή στο μέλλον και πάντως να τους αποφασίσουμε τώρα και να ενημερώσουμε έτσι ώστε να μπορέσει να προβεί σχετικές επενδύσεις η ε, ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικού. Γιατί όσο πιο φιλόδοξοι είναι οι στόχοι, τόσο πιο ε, βέβαιο ότι θα επιτευχθούν. Και επίσης, Πρόεδρε, είμαστε ενώπιον ενός κόσμου διαρκώς μεταλλασσομένου. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τα, στις στις επόμενες δεκαετίες, Κάποιοι θα κερδίσουν, κάποιοι θα χάσουν, ε, κάποιες επιχειρήσεις θα κερδίσουν, κάποιες θα χάσουν, κάποιες ε, χώρες θα κερδίσουν και κάποιες θα χάσουν. Θα είναι κερδισμένες και χαμένες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εάν δεν επενδύσουμε ακόμη περισσότερο και αν δεν αποστείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα, την κατάλληλη δομή για την, ε, αν δεν δείξουμε στην βιομηχανία μας τι είδους δομές θα πρέπει να ακολουθήσει για να βρεθεί με την πλευρά των κερδισμένων, τότε σίγουρα θα είναι από τους χαμένους και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ, Chris Davis, για την παρουσίαση αυτή, την εισήγηση σε μια γενική και πιστεύω ε, καθοριστικής ε, και ενθουσιώδης μας ε, συζήτηση. Είχαμε σκιώδη ηγητέ από την ομάδα μου. Πολλοί είναι συνάδελφοι που επίση έχουν ενδιαφερθεί για αυτόν τον ε, οδικό χάρτη 2050. Και η Λίμνα μου έδωσε την πρόταση με τα επιπλέον ονόματα. Παρακολουθούμε λοιπόν την ε, πορεία του Chris Davis ε, έως την Ολομέλεια. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη έκθεση πρωτοβουλίας, λέει ο κύριος Davis. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα πολλά, πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά ασφαλώς είναι ένα από τα θέματα, μια από τις εκθέσεις που θα προκαλέσουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. γιατί δεν ε, εκπονούμε συχνά εκθέσεις ε, με ορίζοντα 40-50 ετών, μισού αιώνα δηλαδή, τέτοιου είδους οραματισμό δεν έχουμε συνήθως ε, στις εκθέσεις μας, μάλλον προβλήματα στιγμιαία επικαιρότητα ή έστω μέχρι έναν ορίζοντα δεκαετίας καλύπτουμε με τις εκθέσεις μας. Τώρα όμως πάμε μέχρι τα μέσα του αιώνα λίγο πολύ και καλά πιστεύω επέλεξε ο κύριος Ντέιβιτ, όφιλε άλλωστε να επιλέξει αυτόν τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διότι οι δυναμικές ε, στον κόσμο μας, στον τομέα αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλες και χρειάζεται βεβαίως ένα μακροπρόθεσμο σενάριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, τους πολύ φιλόδοξους που θα οδηγήσουν στην μείωση ε, μάλλον στην σταθεροποίηση της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη στους συν 2 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως η, αύξηση, η ανάπτυξη και της οικονομίας ε, συνεπάγεται και αυξανόμενες ανάγκες και κατανάλωση πρώτων υλών, πράγμα το οποίο ίσως σημαίνει επιπλέον αύξηση του βάθρου πάνω στο οποίο έχουμε χτίσει αυτό το σύστημα. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, πιστεύω, βέβαια να προσθέσουμε και τις ΗΠΑ, καλό θα είναι να έχει ένα όραμα για το 2050. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις και ανάγκες για ε, επενδύσεις. Η κύκλη ε, των επενδύσεων ε, για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού είναι δεκαετιών, 40-50 χρόνια κρατάνε αυτά τα εργοστάσια. Είναι επενδύσει μακροπρόθεσμε δηλαδή. Τα εργοστάσια που χτίζονται τώρα θα τα έχουμε και το 2040 να ε, λειτουργούν. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε και ε, εμεί και η κοινωνία μα δηλαδή, αλλά και η βιομηχανία, το τι έρχουμε στο μέλλον, το τι έρχεται στο μέλλον για να μπορεί αναλόγω να προγραμματίσει και να προσαρμοστεί. Σε μια πρώτη συζήτηση που είχε γίνει σχετικά είχαμε πει ότι είναι πολύ πιο φθηνή και αποτελεσματική η πρώιμη, ε, ο πρώιμος σχεδιασμός, η ο, ο πρώιμος προγραμματισμός ε, από τον προγραμματισμό και την υλοποίηση τελευταία στιγμή. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, καταφέρουμε την μεγάλη αλλαγή που θα σημάνει με εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων λίγο πολύ και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο κείμενο της Επιτροπής έχουμε τρεις-τέσσερις μεγάλους τομείς της ενέργειας που θα πρέπει να απελευθερωθεί τελείω από το διοξίδιο του άνθρακα ουσιαστικά, να απαλλαγεί από το διοξίδιο του άνθρακα για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Η βιομηχανία θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό 38 με 83 ε, με 87% περίπου θα πρέπει να απαλλαγεί πάλι από το, τις εκπομπές του άνθρακα. Το ίδιο και για τις μεταφορές, 61 με 64%. Στις δε οικοδομές τα ποσοστά είναι από 88 έως 90%. Άρα όλος ο χώρος κατασκευαστικός, οι οικοδομές δηλαδή, θα πρέπει να απαλλαγούν σχεδόν ολοκληρωτικά από το διοξίδιο του άνθρακα. Μιλάμε δηλαδή για ε, είτε ουδέτερα ενεργειακά, είτε με θετικό ε, ενεργειακό ισοζύγιο ε, σπίτια, κτίρια Το ίδιο και στον τομέα των αυτοκινήτων, των ε, ιδιωτική χρήσεω, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με αυτοκίνητα κινούμενα με υδρογόνο είτε με άλλα καύσιμα. και υπάρχουν και άλλες προτάσεις εκ των οποίων ορισμένες στείνουν προς την πυρηνική ενέργεια τουλάχιστον ε, η οποία τουλάχιστον είναι στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος ε, απαλλαγμένη από εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί στον υπόλοιπο κύκλο της δεν είναι δεδομένο αυτό και άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες τεχνολογίες. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση δηλαδή, μια βιομηχανική επανάσταση που θα έχει και τους νικητές, θα έχει και τους ηττημένους της, ε, που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε φεσή και εξαφάνιση ακόμη ορισμένους κλάδους βιομηχανίας, αλλά θα εξασφαλίσει και την εμφάνιση και επιβίωση και επικράτηση άλλων ε, τομέων της βιομηχανίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν όλους αυτούς τους ε, παράγοντες, όλες αυτές τις πτυχές και εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να τους εξισορροπήσουμε έτσι ώστε να μην είναι πολύ ε, οι χαμένοι και λίγοι νικημένοι ή εκείνοι που έχουν χάσει να έχουν χάσει πολύ. Πρέπει να βρέουμε, δηλαδή έναν τρόπο για, απο... για εξισορρόπηση για αποκατάσταση, για νέα κίνητρα. Χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις για νέα επαγγέλματα, νέες δεξιότητες. Η Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει μεγάλο έργο να επιτελέσει σε σχέση με τις περιφέρειες και τα αστικά μεγάλα κέντρα που χρειάζεται και το ΕΦΤΑ, όπου δισεκατομμύρια των περιφερειακών ταμείων κονδύλια θα πρέπει να βοηθήσουν και θα έχουμε και κάποιους ανθρώπους που θα υποφέρουν τα πάνδυνα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, διότι όλα αυτά θα κοστίσουν χρήματα και όλα θα γίνουν δαπανηρότερα. Το θέμα της παινίας, ενεργειακής παινίας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι σωστό σε αυτό το όραμα για το 2050 να δούμε τα ενδιάμεσα βήματα και να τα περιγράψουμε 2030-2040. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για να, να το κάνουμε αυτό. Έχουμε ένα πλαίσιο μέχρι το 2020 και θα είναι ήδη η χρονική στιγμή να ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον. Πώς θα συνεχίσουμε στο μέλλον. Η Ρωμάνα Τσίζελ είναι εδώ παρούσα που από πλευρά Ήτρε έχει αυτή την έκθεση. Η Ήτρε είναι αρμόδια για την ενεργειακή πολιτική. Χρειαζόμαστε την περιβάλλον και την Ήτρα για αυτό το θέμα. Πρέπει να πούμε και να τοποθετηθούμε ποιος θα είναι ο στόχος, η στοχοθέτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030. Ποιος θα είναι ο στόχος για την αποδοτικότητα εκμετάλλευση ενέργειας μέχρι το 2030. Αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την καλύψει και να την κάνει η και να συνεργαστεί μαζί μας ε, ως προς αυτές τις πτυχέ ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δύο θέματα ακόμα να αναφέρω το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα πρέπει να βοηθήσει. Είναι ισχνά τα κονδύλια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παντού έχουμε κενά και, και ελλείψεις για τις ε, ε εκτός μπροστά στις ακτές μας, ε, τις ε, μονάδες και αλλού λείπουν τα κονδύλια. Και τέλος, τέλος χρειαζόμαστε και τα σωστά μηνύματα που θα δώσουμε όσον αφορά τα κίνητρα και τις τιμές. Με μια τιμή 7 ευρώ, το ανέφερε ο Chris Davis, ή και 16 ευρώ. <coughs> Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες ιδέες που θα δίνουν τα σωστά μηνύματα και που θα βοηθήσουν ως κίνητρα να επιτευχθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Να αναφέρω όμως παρόλα αυτά ότι η διαρροή άνθρακα Carbon Leakage συμφωνώ ότι έχουμε ένα ανταγωνισμό μεταξύ πράσινων τεχνολογιών στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να αναμείνει, να περιμένει η Ευρώπη, θα πρέπει να προχωρήσει προ τα εμπρό. Έχουμε όμω προβλήματα με κάποιου τομεί και η διαρροή άνθρακα, carbon leakage, είναι μέρο αυτή τη προσέγγιση. Αν δεν υπάρξει κοινή κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι, θα πρέπει να υπάρξει ένα αντισταθμιστικό μηχανισμό ή μια αντιστάθμιση συνοριακή. Να μην τιμωρούνται οι δικέ μα βιομηχανίε και άλλοι αθέμητα να αποκομίζουν πλέον ε, πλεονεκτήματα από αυτή την κατάσταση. Έχουμε έναν αρκετά μεγάλο κατάλογο αγορητών. Η Ρωμάνα Γιορντάν Σίσελη θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. έχω έναν άλλο ρόλο σε σχέση με το ψήφισμα για τις κλιματικές αλλαγές πλέον. Διότι εδώ δεν εκπροσωπώ την Επιτροπή Βιομηχανία στην Ήτρα, αλλά είμαι σκιώδη εισηγήτρια για την ίδια την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Κατά τα άλλα, συμφωνώ μαζί σα, Πρόεδρε. Συμφωνώ και με αυτά τα οποία είπε κατά τα άλλα ο εισηγητή, ότι αυτό το έγγραφο, με άλλα λόγια, είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και ιδιαίτερα βλέπω την αναγκαιότητα να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε μετά το 2020 και να δώσουμε <clears throat> μεγαλύτερη προσοχή στην πορεία στο μέλλον. Δεν θέλω να επισέθω υπερβολικά σε λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αναλώσουμε υπερβολικά την ενέργεια. Πρέπει να βρούμε ένα γενικό προσανατολισμό. Και κατά τούτο ελπίζω ότι το έγγραφο το οποίο θα έχουμε στα χέρια μας στο τέλος, θα υποστηριχθεί και μέσα στο πλαίσιο των άλλων εγγράφων που είναι σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς τους στόχους μας μέχρι το 2020 θα θέλαμε να τους επιτύχουμε, να τους υλοποιήσουμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρα προετοίμασε αυτό το έγγραφο. Διότι ο στόχος μας είναι με άλλα λόγια να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο, μια απαιτητική στοχοθέτηση αναβαθμισμένη για τις εκπομπές ρήπων και γι' αυτό από το 2020 και μέχρι το 2050 χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμους στόχους. Στόχος μας τελικά θα είναι μια κοινωνία με χαμηλά επίπεδα άνθρακα. Αυτό σημαίνει μεγάλες επενδύσεις και καινοτομία από πλευράς ε, βιομηχανιών και καινοτομία στις επενδύσεις και σταθεροποίηση που πρέπει να επιτευχθεί. Και για να επιτευχθεί αυτή η σταθεροποίηση χρειαζόμαστε κοινούς ε, και αξιόπιστους ε, στόχους. Και στη συζήτηση για αυτό το έγγραφο δεν θα φανταζόμουν θα έπρεπε να συζητήσουμε αν είναι σωστή η στόχοι μέχρι το 2020 ή όχι. Έχουμε θέσει αυτούς τους στόχους ούτως ή άλλως και πρέπει να τους επιτύχουμε και μακροπρόθεσμα είναι και αναγκαίοι. όλα αυτά όμως πρέπει να διατυπώσουμε το ερώτημα πώς επιθυμούμε να τους υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους χειροπιαστά. Διότι αυτή η χρονική στιγμή είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι αναγκαίο μέχρι το 2030, μέχρι το 2040, μέχρι το 2050 να γίνει όσον αφορά εξειδικευμένους στόχους. Είναι σημαντικό όμως αυτοί οι στόχοι να τεθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές πλαίσιο και να διεθνοποιηθούν, να παγκοσμιοποιηθούν. Η συζήτηση για αυτά τα θέματα σε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να διαρκέσει επαρκέ χρονικό διάστημα ώστε να λάβουμε επαρκώ υπόψη αυτά τα οποία κατά τα τέλη του έτου, σε συνδιάσκεψη για το κλίμα και τι κλιματικέ αλλαγέ θα συζητηθούν. Επίση θα, ήθελα να συζητήσουμε πώ μπορούν οι εκπομπές ρήπων συνολικά να μειωθούν. Μέχρι σήμερα αυτή η συζήτηση χαρακτηριζόταν στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εκπομπές ρήπων μόνο από την επικέντρωση, την εστίαση που είχαμε στην πλευρά της παραγωγής, στην συνιστόσα της παραγωγής. Αν όμως θέλουμε να είμαστε σοβαροί με την αναχέτηση της αύξησης της ε, θερμοκρασίας ε, στον πλανήτη, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να κρίνουμε τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας συνολικά, ποιους στόχους θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και τι θα συμβαίνει σε σχέση με αυτούς τους στόχους ε, και ποιες συνέπειες θα υπάρξουν. Μόνο έτσι μπορούμε ως ε, παγκόσμια κοινότητα να είμαστε αξιόπιστοι και να καταφέρουμε να μειώσουμε και την αύξηση της θερμοκρασίας και την, τις κλιματικές αλλαγές και μόνο τότε θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλη είναι η διαρροή άνθρακα, ποια εμβέλεια έχει. Και γι' αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι σημαντικό να, να υπάρξουν κίνητρα για την ε, βιομηχανία μας, για τις βιομηχανίες μας, να υπάρξουν κίνητρα από τη μια πλευρά έχουμε τη βιομηχανία, από την άλλη πλευρά φυσικά έχουμε και τον ενεργειακό τομέα που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός οπωσδήποτε. Δεν έχουμε μόνο μια παλαιά υποδομή, βιομηχανική υποδομή, αλλά έχουμε και μια ανεπαρκή υποδομή. Εδώ τεράστιες επενδύσεις απαιτούνται για να προχωρήσουμε. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνουν σε μια ανάλυση, γίνεται μια ανάλυση υπό διαφορετικές πτυχές και συνιστώσεις. Αυτό αναφέρθηκε και δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτή η προσέγγιση θα έλεγα είναι καλή. Θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να μετατεθεί, να μεταφερθεί την παγκόσμια κλίμακα στην, ε, μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ε, μείωση των εκπομπών ρήπων. Τις εκπομπές ρήπων δεν θα καταφέρουμε έγκαιρα να τις μειώσουμε αν δεν θα έχουμε μια αντίστοιχη τεχνολογική ανάπτυξη, για να επιτευχθεί αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδος χρειαζόμαστε επενδύσεις. Πρέπει η καινοτομία, η έρευνα και η καινοτομία να προαχθούν και πρέπει αυτοί οι στόχοι με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα να συνδεθούν, πράγμα το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση, υπό ε, σχεδιασμό αυτή τη στιγμή και αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προκατακτικά έγγραφα το φθινόπωρο του έτους εφέτος να τα υποβάλει. Αυτό το έγγραφο Horizon 2020, ο ορίζοντας 2020, πρέπει να είναι προσέγγιση και κίνητρο για μας ώστε να αντανακλώνται τα προβλήματα, τα συνολικά προβλήματα για τις κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά πρέπει να συνδέονται και με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση, το προανέφερα αυτό πιο πριν, είναι για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν επιτρέπεται να αμελήσουμε αυτή την πτυχή. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και τις τρεις πτυχές της αηφορίας ε, στην ανάπτυξη να συλλάβουμε υπόψη την κοινωνική πτυχή, αλλά αφετέρου και την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον, τις περιβαλλοντικές πτυχές. Όλα αυτά πρέπει να τεθούν συνολικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται να αμεληθεί καμία από αυτές τις συνιστώσεις. Κάποιες ερωτήσεις τώρα σε σχέση με την ανάγνωση του εγγράφου όπως ε, ε, είδα κάποια πράγματα, διάβασα και κάποια βιβλία για αυτά τα θέματα και γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα, διαφορετικά μέσα χρηματοοικονομικά με τα οποία θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ε, υπέρ της προστασίας του κλίματος. Τώρα για το ερώτημα ποιο μέσο θα πρέπει να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί. Εδώ έχουμε και την συνάρτηση με τις διαφορετικές τιμές για την, ε, το αντίτιμο του διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ έχουμε διαφορετικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθούν και αυτά υπόψη. Βλέπω να απουσιάζει, να απουσιάζει μια εκτίμηση πώς και πόσο θα στοιχήσει στον μέσο πολίτη στους φορολογούμενους αυτή η μείωση των εκπομπών ρήπων. Συμφωνώ με, κατά τα άλλα με αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν. Εμείς θα πρέπει τεχνολογικά όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι και αμερόληπτοι να είμαστε. Δεν επιτρέπεται εκ προημίου τη τιμή, το κόστος ε, τη τεχνολογίας να τα προκαθορίσουμε δεσμευτικά. Εδώ τίθεται ωστόσο από την άλλη πλευρά ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την πυρηνική ενέργεια μόνο η ε, σύνδεξη, η σχάση με συγχωρείτε αναφέρεται και θα πρέπει να δούμε ότι σε σχέση μέχρι το 2020 για την πτυχή αυτή που πρέπει να λάβουμε υπόψη, θα ήθελα να γνωρίζω πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στου υπολογισμού από πλευρά τη, τη συνιστόσα τη πυρηνική ενέργεια και το τμήμα τη πυρηνική ενέργεια ε, ω συνιστόσα τα εκτιμά ω στοιχεία. Νομίζω η κύρια εστίαση Παράλληλα με την πυρηνική ατομική ενέργεια πρέπει να ευρίσκεται η επικέντρωσή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξίσου. Θεωρώ ότι το έγγραφο αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ καλό. Θα έπρεπε να προ προσπαθήσουμε, πιστεύω, αν είναι δυνατόν να βρούμε τα πιο εξειδικευμένα και σωστά μέτρα. Είναι σωστή η προσέγγιση και το προανέφερα. Πρέπει ωστόσο να μην κατακαιρματιστούμε στις λεπτομέρειες και χάσουμε τη σωστή πορεία, την σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να εγκρίνουμε τις προτάσεις στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτευχθεί μεγάλη συνένεση. Είναι σημαντική πρωτοβουλία του εισηγητή αυτό το έγγραφο να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία άσκησης θετικής πίεσης από το Ευρωκοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουμε όμως ρεαλιστές, ρεαλιστές με ρεαλιστικό πνεύμα να τα τα δούμε αυτά είχα να πω ευχαριστώ. Um, Σε ευχαριστούμε πολύ Ρωμάνα. Ήμουν κακό παράδειγμα. Δέκα λεπτά που υπήρξε η παρέμβαση. Οι συντονιστές θα πρέπει να ε, ε, είναι πιο σύντομοι, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος ε, κατάλογος αγοριτών ή δυνατόν να είσαστε συντομότεροι και στο τέλος θα καταφέρουμε να, να καλύψουμε τα θέματα της έκθεσης αυτής. Αν ξεκινήσουμε έτσι τότε και τον δικό σας χρόνο σήμερα το πρωί θα πρέπει να τον συνυπολογίσουμε πρόεδρε που μιλούσατε και είχατε την αποκλειστικότητα στην παρέμβασή σας. Θα είμαι σύντομο για αυτό το θέμα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι κάθε, κάθε φορά όταν συζητάμε τον, τον οδικό χάρτη για το 2050 όλοι φαίνεται να συμφωνούν διότι φαίνεται ότι είναι ένα μια μεγάλη πορεία, μακρά πορεία μέχρι το 2050 και μπορεί, μπορεί να λένε έτσι όλοι ότι συμφωνούμε για τους στόχους του 2050. Όμως όταν συζητάμε το θέμα του οδικού χάρτη για το 2050 είναι το να απαιτείται και να καλυφθεί η πλήρης μετατροπή της οικονομίας μας που πρέπει σε διαφορετικά επίπεδα να ξεκινήσουν κάποιοι να ξεκινήσουν ήδη αύριο ή και μεθαύριο όμως το 2050 βρίσκεται πολύ πιο κοντά από ό,τι υπολογίζουμε και γι' αυτό χαίρομαι για το ότι ο εισηγητής τονίζει αυτό το, το, το θέμα στο έγγραφο εργασίας του. Νομίζω σε σχέση με τις επικρίσεις για τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφές είναι ότι έχουν αναφέρει προημίου ότι πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος ε, μεταβατική περίοδος όσον αφορά μια χαμηλή εκπομπές ε, ρήπων ε, οικονομία και όταν κάνουν λόγο για τα ορόσημα milestones όπως και να το αποκαλέσετε, ορόσημα, στόχους, αυτά που θα γίνουν σε περίοδο 40 ετών, θα έχουμε μια μείωση 40% και τα τελευταία χρόνια θα έχουμε άλλη μια κατά 40% μείωση. 80% μείωση συνολικά. Σε 40 χρόνια 40% για άλλα 20 χρόνια, στα επόμενα άλλα 20 χρόνια, πάλι για άλλη μια φορά 40% μείωση και βλέπουμε έτσι ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά την μείωση ε, των εκπομπών ρήπων, να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν είναι καθόλου γραμμική η εξέλιξη και η ανάπτυξη και αυτό δεν είναι καλό γιατί κάποιοι τομείς πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν ώστε να μπορέσουν άλλοι τομείς να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές ακόμα περισσότερο στη συνέχεια, υστερότερα. Αν πάμε γραμμικά από το 1990 στο ε, το 2040 ε, 10% ανά δεκαετία που δείχνει μέχρι το 2020 κατά 30% μείωση είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ως Κοινοβούλιο την τομεακή προσέγγιση συζητώντας αυτόν τον οδικό χάρτη. Για παράδειγμα αναφέρθηκε επίσης από τον κύριο Ντέβις και αν δείτε τη μεταβατική περίοδο για την οικονομία ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο πιο κρίσιμος τομέας που πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα. Αν δεν αλλάξει δραστικά τις δομές του στο άμεσο μέλλον αυτός ο τομέας, ε, τότε μπορούμε να αναμείνουμε σε σχέση με τους άλλους τομείς που εξαρτώνται από αυτόν τον τομέα για να δούμε το τι θα μπορέσει να γίνει. Και αυτό τονίζει, μας κάνει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο την ανάγκη ο τομέας παραγωγής, ο κλάδος παραγωγής ενέργειας να κινητοποιηθεί και να κινηθεί πρώτος. Μιλάμε πάντα για χαμολές εκπομπές ρήπων τι σε, σε άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό. Ένας τελείως διαφορετικό, ένα τελείως διαφορετικό τομέα παραγωγής και στη μεταβατική περίοδο όσον αφορά την σύνδεση με το φυσικό αέριο τελείως διαφορετικό τομέα από εκείνον που ε, ε, είχε αποκλειστική εξάρτηση από τον άνθρακα στο παρελθόν και μετά είχε και μετάθεση στην πυρηνική ενέργεια. Κάνουμε λόγο για συζητάμε ένα τελείως διαφορετικό τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αν θέλετε μακροπρόθεσμα να πετύχετε κάποιους στόχους οι αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα και να μην συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως το παρελθόν και να συνεχίσουμε την ε, παρελθούσα ας πούμε δράση και στο μέλλον με την χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αμέσως στη συνέχεια είναι η αποτελεσματικότητα και αυτό όλο και περισσότερο πρέπει να τονίζεται. Αν δείτε όλες τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και ξέρω ότι η κυρία Τζόρνταν ζητεί να υπάρξουν περισσότερες μελέτες αλλά υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν ήδη συνταχθεί. Αν τις δείτε και τις διαβάσετε όλες με σαφήνεια κάθετα λένε ότι αν θέλετε να κινητοποιηθείτε και να καταφέρετε να έχετε το δυνατόν πιο προσιτές φθηνές τιμές, τότε πρέπει να διασφαλίσετε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Διότι όσο λιγότερο σπαταλάμε και ε, καταναλώνουμε ενέργεια περίτα, τόσο ε, θα είναι αναγκαίο να πούμε ότι όσο μειώνεται αυτή η διασπάθηση ενέργειας θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την κοινοβουλευτική μας επιτροπή σε στενή συνεργασία βέβαια με την Επιτροπή Βιομηχανίας, την Επιτροπή Ήτρε. Το σημαντικότερο είναι στην έκθεσή μας αυτή να αναφέρουμε άμεσες δράσεις, ε, δραστηριοποίηση άμεση που πρέπει να αναλυφθεί. Είναι ωραίο να μιλάμε για μακροπρόθεσμους στόχους και μακροπρόθεσμους χρονορίζοντες, αλλά πρέπει να επιτευχθούν άμεση δραστηριοποίηση και αποτελεσματικότητα για να είμαστε στο τέλος να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Κάνουμε λόγο για τη μελλοντική οικονομία, την οικονομία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι σαφές ότι πρόκειται για τη μελλοντική οικονομία και πρέπει να υπάρχουν χειροπιαστές απλές ε, δράσεις, μετάθεση που μεταφορά του τομέα παραγωγής ενέργειας, μετά επενδύσεις στον τομέα μεταφορών που είναι ένας πιο δύσκολος τομέας, δυσχερέστερος τομέας που πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά την οικονομία, κάτι πρέπει να γίνει παραπάνω για τις μεταφορές και να διασφαλίσουμε ότι τα κίνητρα από πλευράς τιμών θα διασφαλιστούν ώστε να υπάρχουν σωστά κίνητρα που θα δοθούν στις βιομηχανίες ώστε να δράσουν με το σωστό τρόπο και μετά καταλήγουμε στο χειροπιαστό σύστημα της ε, εμπορίας εκπομπών ρήπων, ITS. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε να το ξαναδούμε για να υπάρξουν οι σωστές τιμές κίνητρα, να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα με τη σωστή αλληλουχία και σειρά. Και γι' αυτό για τον κύριο Ντέβις θα ήθελα να πω ότι δεν θα καταλήξει η ελπίζω η έκθεση του κύριου Ντέβις όπως συνέβη με τη δική μου έκθεση, γιατί καθώς προχωρά ο χρόνος όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να υπάρξουν καλύτερα επίπεδα τιμών και για την ε, εταιρεία Shell για παράδειγμα που αναμένει να δει τι θα πράξει ώστε να κινητοποιηθεί με το σωστό τρόπο προς τις σωστές κατευθύνσεις και να έχουμε και ε, άμεση δράση, δραστηριοποίηση και όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο ενός ε, ευρύτερου χρονοορίζοντα. Ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υποστηριχθεί και να προχωρήσει η έκθεση. Σας ευχαριστώ και είσαστε προπομπός ε, στο να προλιάνετε το έδαφος για τους επόμενους αγορητές για την έκθεση Davis. Μπάρμπαρα Ντεμπρόιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με το υπόθηκαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, και ενδιάμεσοι στόχοι και μακροπρόθεσμοι. Επίσης, θα πρέπει πιστεύω να υπάρχουν ε, σαφείς θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής ιδέα των βημάτων που θα πραγματοποιήσουμε. Επίσης, σε σχέση με τα όσα σήμερα ε, συζητούμε, δηλαδή του στόχους που έχουμε για το 2020, πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε κάποιες ιδέες. Δεν πρέπει να καταλήψουμε το 30% ως ε, πρόθεση. Τι έχουμε πει, είναι και πολύ σημαντικό. Και έχουμε πει επίσης ότι θα πρέπει και ο κλάδος να γνωρίζει τι βρίσκεται στο μέλλον, στον ορίζοντα. Το είπε και ο Chris Davis. Πρέπει να ορίσουμε δηλαδή στόχους, πρακτικούς, μέσο και μακροπρόθεσμα για να γνωρίσει ο κλάδος που θα επενδύσει. Και αν δεν το πράξουμε αυτό, δεν θα γίνει η δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να γίνει. και δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Το θέμα λοιπόν για μένα δεν είναι το αν μπορούμε οικονομικά να αντέξουμε αυτά τα βήματα, όπως ακούστηκε, αλλά το αν μπορούμε να αντέξουμε την μη πραγματοποίηση αυτών των βημάτων. Γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε το κεφάλι στην άμμο, να αφήσουμε τους όλους να μας ξεπεράσουν και όταν έρθει η ώρα να υποχρεωθούμε να εισαγάγουμε ιδιαίτερως από τους άλλους την τεχνολογία που θα χρειαζόμαστε, γιατί θα τη χρειαστούμε τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο τις ε, ε, τεχνολογίες, την καινοτομία που θα χρειαστούν, αλλά και θετικά βήματα, τις θετικές συνέπειες κάποιων μεμονωμένων ενδεχομένω ε, βημάτων εφόσον δεν υπάρξει γενικότερη συμφωνία. Εγώ από τη δική μου δηλαδή την ε, ε, εκλογική περιφέρεια είδα ένα ναυπηγείο το οποίο το ένα χρόνο, μετά τον άλλον είχε όλο και λιγότερη δουλειά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι το εγκατέλειπαν ε, και τελικά αναγκάστηκε να αναπροσαρμοστεί στις ανανεώσιμες, αναγκάστηκε να κοιτάξει την τεχνολογία των κυμάτων, της ενέργειας από κύματα δηλαδή, αυτό είναι θετικό. Αν πραγματοποιήσουμε δηλαδή σωστά βήματα, δεν είναι απαραίτητο να υποφέρει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα υπάρχουν κερδισμένοι και ηττημένοι, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κερδίσει ο ένα τομέα και να χάσει ο άλλο. Μπορεί μέσα στον ίδιο τομέα κάποιο να κερδίζει και να βοηθάει αυτόν το ο οποίο έχει λιγότερο καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να αποστείλουμε. Η δε πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη και σε αυτό δεν υποστηρίζω την ιδέα Επίσης, συμφωνώ με τις προτάσεις για την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας. Πρέπει, πιστεύω, να καταστήσουμε απόλυτα σαφές το πόσο πολύ συμβάλλει στην επιτεύξη των στόχων η ε, η επιλογή αυτή. Και δεν μπορούμε να έχουμε οδικό χάρτη αν δεν ξέρουμε ξεκάθαρα τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Επίσης, δράσεις άμεσες, πολύ σημαντικές με τα όσα είπε και ο κύριος Ντέβιτ, αλλά και εσείς κύριε Πρόεδρος είπα γνώμη στο παρελθόν, ανάγκη για επενδύσεις στον χώρο των μεταφορών, με τεράστια σημασία, εάν θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα, αν θέλουμε να στραφούμε προς τις επενδύσεις, την κοινοτομία, την έρευνα. Και εν τέλει, Πρόεδρε, Έχει υπάρξει όντω πρόοδος με το έγγραφο εργασίας το οποίο δίνει στο Κοινοβούλιο όραμα για το μέλλον. Ναι. Από την άλλη όμως θα πρέπει όχι μόνο να ευχαριστήσουμε τον Chris Davis αλλά και να ορίσουμε τι είδους δράσεις θέλουμε μέσα στο σχέδιο έκθεσης, συγκεκριμένες προτάσεις για τους στόχους για την αποτελεσματικότητα της χρήση ενέργειας, τις επιλογές για τη μετάβαση στις ενεργειακές μας ανάγκες, για την απουσία backloading και επίσης για τις επενδύσεις που θέλουμε και είναι υποχρεωτικό να κάνουμε έτσι ώστε να αποστείλουμε και τα κατάλληλα μηνύματα στον κλάδο. Μηνύματα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξουν εξελίξεις και θα τις στηρίξουμε στις προσπαθίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχήν στους, ε, στους ε, πράσινους συναδέλφους ότι μιλάνε, μιλάνε καλά αλλά οι πράξη τους δεν τους ακολουθούν. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε εμεί ε, αυτό το μπουκάλι νερό γεμάτο με διοξίδιο του άνθρακος. Κάποιος θα άνοιγε το μπουκάλι και θα πεθαίναμε όλοι. Κάποτε ένας καταστροφιστής ε, διακήρυσε στη μέση του Central Park ε, ότι κάποιοι ότι σε δύο-τρία χρόνια θα, θα, θα, θα, σηκουνών, ανέβαινε το επίπεδο ε, της ε, θάλασσας και θα πνιγόντουσαν όλοι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι τελικά ένα έγγραφο πάρα πολύ ωραίο για, μια, για ένα συλλαλητήριο, αλλά όχι για μια κοινοβουλευτική επιτροπή μιλάει για θέματα τα οποία με τίποτα δεν μπορούμε να συμμεριστούμε. Εντάξει, σύμφωνοι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αλλαγές του κλίματος, αλλά πρέπει να γίνει συνολικά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά αν κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς, ε, απλώς βγάζοντας ε, τις ενεργοβόρες, ε, τα ενεργοβόρα εργοστάσια από την Ευρώπη και τα πάμε αλλού. Διότι η ρήπανση είναι ε, παγκόσμια, είναι συνολική. Άμα παίρνουμε εμείς το εργοστάσιο από την Ευρώπη και το πάμε στην Κίνα, η ρήπανση δεν αλλάζει σε τίποτα. Ή εμείς ε, θα είμαστε σε θέση ως Ευρώπη να πιέσουμε ε, ώστε οι διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν στον Τάρμαν τον Δεκέμβριο θα επιβάλλουμε, θα επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες που ρηπαίνουν να μετριάσουν τις εκπομπές τους ή να έχουμε το κουράγιο να υποβάλουμε δασμούς στα προϊόντα των χωρών που ρηπαίνουν και που τα εισάγουμε εμείς στην Ευρώπη. Διότι εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τελικά ότι θα κλείσουμε τα εργοστάσια μας στην Ευρώπη πιστεύοντας ότι κάτι κάνουμε όταν το εργοστάσιο από την Ευρώπη μετά μεταφέρεται στην Κίνα αύξηση διοξιδίου του άνθρακος αυτό το σημείο ελέγχου της ε, νήσου Γουάι. Λοιπόν, ε, γιατί δεν μου το αποδεικνύετε εσείς, ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυτές τις τεράστιες εκρήξεις των ηφαιστείων λίγους μήνες πριν από τις ε, μετρήσεις που ρηπαίνουν σε τεράστιο βαθμό την ατμόσφαιρα. Ελάτε να μου αποδείξετε λοιπόν ότι αυτή δεν ήταν η αιτία και τότε να το συζητήσουμε. Αλλά να μου πείτε εσείς ότι μέχρι το 2050 θα μειώσουμε σε τόσο μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές είναι πραγματικά ουτοπία σίγουρα. Θα ανακαλύψουμε κάποια στιγμή το αυτοκίνητο που λειτουργεί με υδρογόνο, αλλά θα ήταν μια τεράστια καινοτομία αυτή. Αν εμείς ε, προωθήσουμε την ιδέα να χρηματοδοτήσουμε άφθονα την ε, έρευνα, τότε να, θα καταφέρναμε να είχαμε εμείς ε, τέτοιου είδους ε, αυτοκίνητα για να μειώσουμε τη ρήπανση, μπορεί να το καταφέρναμε. Αλλά το να λέμε εμείς σήμερα στα εργοστάσια μας ότι θα πρέπει να μειώσουν μέχρι το 2050 κατά 80-90% τις εκπομπές τους. Είναι σαν να λέμε στο ευρωπαϊκό εργοστάσιο δεν επενδύεις πια στην Ευρώπη, κλείς το μαγαζί και πήγαινε σε μία τρίτη χώρα, κάνε την επένδυσή σου και σκασίλα σου το περιβάλλον, λέει ο μιλητής. Αυτό είναι κάτι που ένας πολιτικός, ένας νομοθέτης δεν θα έπρεπε να το κάνει και μετά. Μα πραγματικά δηλαδή είναι τρομερό. Πώς μπορεί κανείς να γράφει στην έκθεση ότι δεν υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοκίνητοβιομηχανία, όταν όλες οι οικονομικές εφημερίδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο λένε ότι υπάρχει μία τεράστια μείωση των κερδών της αυτοκίνητοβιομηχανίας. Αυξήθηκε το κόστος, μειώθηκαν οι πωλήσει. Μην λέτε εδώ ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις, σε πραγματικά. Αυτό σημαίνει ότι ο εισηγητής δεν άνοιξε ποτέ του μια οικονομική εφημερίδα. Διότι δεν γνωρίζει προφανώς ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τεράστια κρίση σήμερα στον τομέα της αυτοκίνητοβιομηχανίας και πολλές ε, μπορεί να αποφασίσουν να κλείσουν. Εξάλλου πολλές ήδη έχουν μετατοπίσει τις εγκαταστάσεις τους και άλλες μπορούν να κλείσουν ή να και να μετατοπίσουν. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη ε, κατά τη γνώμη μου είμαι αντίθετος σε αυτήν εδώ τη διακήρυξη ότι η Ευρώπη θα πρέπει αυτόνομα να μειώσει τις, ε, εκπομπές. Με αυτό το έγγραφο τελικά δεν είναι κοινοβουλευτική έκθεση, ε, προκήρυξη συλλαλητηρίου είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώση για τις ξεκάθαρες δηλώσεις σας, των πεπιθήσεών σας. Μάριο, Πρέιο, Όλγα Κράμερ, Χόλγαρτ Κράμερ. Θέλετε και εσείς να λάβετε το λόγο έτσι, Να Ας ακούσουμε τον κύριο Κράμερ πρώτα, πρέπει να πάει στη 4 άλλη επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο πολύ φιλικό και ευχαριστώ. Μια συζήτηση πιστεύω για ένα έγγραφο εργασίας σίγουρα είναι σκόπιμο στοιχείο να διεξαχθεί μια συζήτηση σε, ε, επί των θεμελίων, ε, στη σωστή βάση δεν ξέρω αν είναι η σωστή σκηνή, τα πράγματα λιγότερο συναισθηματικά, λιγότερο ιδεολογικά να τα συζητήσουμε από ό,τι έγινε μέχρι σήμερα. Εγώ προσωπικά, όπω όλοι γνωρίζετε, προέρχομαι από την πρώην Ανατολική Λαοκρατική Γερμανία. Εκεί μεγάλωσα. Και μετά την αποτυχία του κράτους εκεί έχω τεράστιε επιφυλάξει έναντι όλων των μεγαλόπνων πολιτικών σχεδίων που συντάσσονται και συγκροτούνται, ιδιαίτερα έναντι μεγαλόπνοων χρονικών οριζόντων. Γιατί, πολύ απλά, διότι μέχρι σήμερα πάντα αποτύχαναν και η πραγματικότητα τα ισοπαίδωνε. Και γι' αυτό κάποια στοιχεία και ίσως ε, θα, ε, και πρέπει να το δούμε αυτό, το μεγαλοσοσιαλιστικό ε, πρόγραμμα για την Σοβιετική Ένωση. Ο Στάλιν είχε την έμπνευση να λιώσει τους πάγους στην Σιβηρία θα μπορούσε έλεγε να αλλάξει το, τις κλιματικές ε, συνθήκες ώστε να λιώσουν οι πάγοι της ε, Σιβηρίας σήμερα είναι κάπως αξιοπρόσεκτο, κάπως αξιοπερίεργο αυτό διότι γνωρίζουμε όλοι ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Όλα τίθεται υπό επί των θεμελίων του ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιεί το. Και η ευρεία συνένεση όσον αφορά τον Κόνραντ Άντενάουαρ και τον Βίλι Μπράντα από την πυρηνική ενέργεια θα προερχόταν σε σχέση με την ε, Δυτική Γερμανία. Ξέρουμε ε, σε σχέση με το τι συνέβη στην ε, πρώην Δυτική Γερμανία και ότι σήμερα η Γερμανία έχει αποφασίσει να πάψει να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια πια. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για, την, για τέτοια μεγαλόπνοα σε χρονορίζοντα σχέδια είναι σαν να έχουμε μονοπόλιο των γνώσεων και της σκέψης είμαστε ε, αλαζόνες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε τέτοιο ε, χρόνο Κανένας πριν από μερικές δεκαετίες δεν σκεφτόταν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, ενέργειας στο διαδίκτυο και άλλα. Να μην έχουμε τέτοιου είδους χήμερες, γιατί η πραγματικότητα ίδια ισοπεδώνει τέτοιου είδους χήμερες, όπως και τα σχέδια του Στάλιν που οι μετέπειτα γενές ε, σκεφτόντουσαν μα τι είχαν πια υπόψη τους ε, αυτοί οι ηγέτες εντός εισαγωγικών. Και όταν έχουμε μπροστά μας το έγγραφο του Chris Davis και τις προτάσεις. Επιτέλους ήρθε η χρονική στιγμή εμείς οι ίδιοι να διαρωτηθούμε. Τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε όλα και είναι πλέον καθοριστικά και τελεσίδικα όλα αυτά όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Εδώ και χρόνια, χρόνια αναφερόμαστε στο IPCC, το Συμβούλιο για τις Κλιματικές Αλλαγές έχω την εντύπωση ότι είναι σκόπιμο το ερώτημα. Να ρωτήσουμε μόνο, δεν έχω κάποιους ισχυρισμού ή επιχειρήματα. Ήταν πραγματικά αντικειμενικές επιστημονικές γνώσεις αυτές στις οποίες βασιζόντουσαν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι επιστήμονες που λένε ότι δεν εισακούστηκα διότι είχα διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν διαφορετικά συμπεράσματα τα οποία συντάχθηκαν χωρίς να είμαστε αρκετά αυστηροί όσον αφορά την εξέταση και αξιολόγησή τους από ισότιμους επιστήμονες από μια ομάδα επαϊόντων. Και γίνεται εδώ και λόγος για το ε, UK ε, Harley Center για την αύξηση της θερμοκρασίας ε, του ε, παγκόσμιου κλίματος θα μπορούσα εξίσου να αναφερθώ στο ε, Ίδρυμα Τεχνολογιών, Institute of Technologies, που ξεκινά από τελείως διαφορετικές ε, υποθέσεις εργασίας και καταλήγει σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Θα ήθελα και σε σχέση με την, τους Γερμανούς επιστήμονες να αναφέρω έναν Γερμανό επιστήμονα, ο οποίος λέει ότι εκπλήσεται από τον πολιτικό ζήλο κάποιων συναδέρφων του, που θυμίζει και κάπως τον Μακάθη. Εδώ τι πρόκειται για επιστήμη αποκλειστικά ή για την επιβεβαίωση κάποιων πραγμάτων που πολιτικά κάποιοι τα ήθελαν ώστε να κινητοποιηθεί μια τέτοια δυναμική σε σχέση με τους πολίτες ώστε να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις των πραγμάτων. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που ίσως μας πείθουν να πούμε ότι ίσως δεν τα ξέρουμε όλα και υπάρχουν πράγματα που πρέπει ακόμα να μάθουμε και ολοκληρώνω λέγοντας θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο υπόλοιπο κόσμος τη δική μας στρατηγική δεν την ακόμα δεν έχει πιστεί ο υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχουμε καμιά ευκαιρία να επιτύχουμε μια διεθνή συμφωνία για όλου αυτού του στόχου όπω εμεί παρουσιάζουμε τι θέσει μα και αυτό επειδή έχουμε διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικέ θέσει. Όχι να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια συμφωνία, αλλά να προβληματιστούμε να δούμε αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική στρατηγική. Παράδειγμα, με δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την έρευνα σε παγκόσμια κλίμακα Λαμβάνοντα υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα σε άλλε ε, περιφέρειες, περιοχέ του κόσμου και την ανάγκη του να υπάρξει προσαρμογή σε όλε αυτέ τι εξελίξει. Ευχαριστώ επειδή δεν μπορεί κανεί να πει τίποτα ε, περισσότερο πλέον σε αυτή την Επιτροπή και πρέπει να αποχωρήσει, γι' αυτό του δώσαμε δύο λεπτά. Ακούσατε όλοι τι είπε ο Χόλγκα Κράμερ και περνάμε στον εισηγητή τη Ήτρα, Ήτρε, Μάριο Πυρίλιο για αυτό το θέμα. Ο κύριο Πυρίλιο έχει τον λόγο. Μάριο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντέιβις ε, για όλα όσα αναφέρει στο κείμενό του αλλά και γιατί διαφωτίζει το τι εμπλέκουν οι στόχοι της, ε, του οδικού χάρτη στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα στην Ένεση. Είναι πολλά και ετερογενή τα στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Ντέιβις και η συζήτηση θα είναι πολύ ζωντανή και δύσκολη. Διότι εδώ θέλουμε εμείς να κάνουμε σύνθετες επιλογές που εμπλέκουν και την Επιτροπή μας και την Ήτρε. Ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συνένεση όταν θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Η roadmap συλλέγει όλες τις ανησυχίες, δηλαδή τις κλιματικές αλλαγές, τονίζει την σχέση της συγκρέντρωσης ε, διοξιδίου του άνθρακος και αύξησης ε, της θερμοκρασίας, έστω και αν δεν υπάρχει ομόφωνη επιστημονική συνένεση γι' αυτό. Θέλει λοιπόν να φτάσουμε σε μια κοινωνία με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών και να κρατήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία χωρίς παραπάνω μειώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές, αποτελεσματικές δράσεις βράχη πρόθεσμα, χρειάζονται όμως και σύνολοι κα όραματα με ρεαλιστικά εφαρμοστικά μέτρα που θα πρέπει να ξεκινήσουμε το νωρίτερο το δυνατό με πλονεκτήματα όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την απασχόληση και για την οικονομία. Έχουμε πάρα πολλούς ε, ε, δρόμους μπροστά μας και πρέπει να τους ακολουθήσουμε όλους μαζί διότι καμία μεμονωμένη δράση θα οδηγούσε σε μείωση εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος διατηρώντας ταυτόχρονα και ανταγωνιστική την οικονομία. Κατά τη γνώμη μου έχουμε τρία βασικά πράγματα. Έχουμε αυτάρκεια έρευνα, ενεργειακή αυτάρκεια έρευνα και μείωση σημαντική των εκπομπών. Να σας θυμίσω, ξεκινώντας από το τελευταίο. Ο έλεγχος των κλιματικών αλλαγών είναι ένα παγκόσμιο αγαθό για το παγκόσμιο όφελος. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συλλογική μείωση. Η Ευρώπη συμβάλλει με το 10% των παγκοσμίων εκπομπών. Θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα της Ένωσης να, να εμπλέξει και τις μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες εκτός Ένωσης, μειώνοντας τις εκπομπές. Η έρευνα είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές. Θα πρέπει να ενταχθούν στο Horizon 2020, στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, για να βρούμε λύσεις όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την απόδοση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας όπως επίσης και να βρεθεί λύση για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος. Τώρα, το πιο επίγον, αυτάρκεια, ενεργειακή αυτάρκεια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το 20% ε, περικοπών που ορίζει η Ατζέντα 2020 δεν θα, φτάσει, δεν, θα, δεν θα επιτευχθεί εύκολα. Πρέπει εμείς να προχωρήσουμε στην αυτάρκεια ενεργειακή αυτάρχεια των κτηρίων με επενδύσεις στην, στο rating και στην ευφύ οικοδόμηση. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα στοιχεία που πρέπει να προωθήσουμε κατά την πρώτη περίοδο. Ευχαριστώ Μάριο Πυρίλο. Για τη συμβολή σου από την πλευρά της ε, Επιτροπής Ήτρα και συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Chris. Πολύ καλή δουλειά. Οι περισσότερε χώρες έχουν ε, Ακαδημία Επιστημών. Εθνική. Περισσότερες. Και ουδεμία Ακαδημία Επιστημών έχει εκφράσει αμφιβολίες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν έχει αμφισβητήσει την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή ως αποτέλεσμα της δράσης του ανθρώπου. Επομένως, το να συζητά κανείς, συζητεί κανείς εάν το έχει προκαλέσει, προκαλέσει ο άνθρωπος το ζήτημα αυτό, είναι ήδη, νομίζω, λάθος τοποθέτηση. Να σας το πω διαφορετικά. Αν πάτε στο γιατρό γιατί έχετε στη θάχη και σας πει είναι πολύ σοβαρό πρέπει να κάνετε, να λάβετε αυτή και αυτή την αγωγή και φεύγοντα, αποφασίσετε ότι δεν σε εμπιστεύσει το γιατρό αυτό και πάτε σε ένα δεύτερο γιατρό και σα πει το ίδιο, την ίδια αγωγή και ο τρίτο και ο τέταρτο και ο εκατοστό ακόμη. Ε, δεν θα την πάρετε τελικά την αγωγή, δεν θα πρέπει να την πάρετε. Το να αμφισβητεί κανεί δηλαδή αυτή την διάγνωση είναι γελίο ή μη τι άλλο. Βλέπω όμω δυστυχώ ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή που ακόμη το αμφισβητούν. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει, στον σκόπο μου να κοιτάξουμε πω συμφωνήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Αναμφισβήτητο. Κάτι στο οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, ακόμη και αν δεν εντοπίζει κανεί το πρόβλημα στην ε, κλιματική αλλαγή, ή αν δεν θεωρεί ότι την προξενεί ο άνθρωπο στην κλιματική αλλαγή, μπορούμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω, στο ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, μόνο να αυξηθούν. Μπορούν, αν συνεχίσει με την ανάπτυξη του 8% που έχει η Κίνα στην παραγωγή της, το 2030 θα χρησιμοποιεί 99 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα η Κίνα. Ολόκληρος ο κόσμος τώρα χρειάζεται 84 εκατομμύρια βαρέλια. Όλος ο κόσμος, όλες οι χώρες του κόσμου. Αυτό λοιπόν μας δείχνει νομίζω κατά τον τρόπο ότι θα ανέβουν στα ύψη τιμές του πετρελαίου. Άρα λοιπόν ακόμη και αν δεν το βλέπετε σαν πρόβλημα του, του περιβάλλοντος αυτό, οπωσδήποτε θα πρέπει τουλάχιστον να συμφωνείτε ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων και ότι σε μειονεκτική θέση θα βρεθεί η Ευρώπη από ολόκληρο τον κόσμο. Εχθές μόλις ε, εγκρίθηκε, ε, δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση στη Δανία η οποία κατέθεσε το πρόγραμμά της, έδωσε τις ε, προτάσεις της για τη διακυβέρνηση με πρόταση να μειώσει τις εκπομπές του του άνθρακα για το 2020 κατά 40% ή η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά το 20% να προέρχεται από την αιωλική ενέργεια και το 45% η ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό δηλαδή αλλά και θέρμανση να προέρχεται στο 50% από τις ανανεώσιμες πηγές, το δε 2050 ε, να έχουμε φτάσει στο 100% ουδέτερης, ουδέτερου σεζυγίου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να δούμε και άλλες χώρες ε, στην επιλογή αυτή, να μπορέσουμε δηλαδή την ε, απόφαση να την μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος, ευχάριστα από την Κοπενχάγη, πολύ καλά. Είχαμε και κακά. Ναι, από τη χάρη γυρνάει και τα καλά. Αυτό τουλάχιστον μας ευχαριστεί. Ο Καλ Χάινς Φλόρενς. Και εγώ πάντα χαίρομαι όταν ακούω καλά μαντάτα από τα κράτη-μέλη. Θετικές ειδήσει. Διότι δυστυχώς σε αυτό το ζήτημα δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Και γι' αυτό επιμένω και λέω ότι πρέπει σε βάθος να δούμε όλα σωστά τα εγκρίναμε και τα αποφασίσαμε και τι υλοποιήσαμε στις χώρες μας. Και μπορούμε αμέσω τότε στη Γερμανία να δούμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και διαφορές. Και δεν ανήκω σε εκείνους που παίζουν με αριθμητικά μεγέθη και ρίχνουν κάποια στοιχεία αριθμητικών μεγεθών. Υπάρχουν κάποια στοιχεία επί των οποίων μπορώ να πω ότι χρειαζόμαστε τα αριθμητικά στοιχεία ουσιαστικά και τις τις διορίες, τις προθεσμίες. Γιατί σε σχέση με τους βιομηχάνους, όποιος θέλει να σχεδιάσει και να προγραμματίσει πρέπει να έχει στοιχεία για την δράση και τη βιομηχανία του. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ορθοποδήσει και να προχωρήσει κανείς. Χρειαζόμαστε ένα μέσο, ας το πω έτσι, πρόγραμμα σε σχέση με, το φυσικό αέριο και μετά από 40 χρόνια ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό αυτές ε, οι μακρές περίοδοι είναι σωστή προσέγγιση. Και για τον συνάδελφο Κράμερ, τα παίρνω έτσι ε, εναλλάξει σταχυολογώ από τις παρεμβάσεις που έγιναν. Για τον κύριο Χόγκερ Κράμερ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τα άκουσα αυτά κάποιες φορές. Ήμουν και εισηγητής και αν θέλετε εδώ να έχω και προσωπική τοποθέτηση, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι τοποθετούνται κατά των κλιματικών αλλαγών και δεν είναι παρόντες ας πούμε στην όλη συζήτηση και είναι δημοφιλής με τέτοιες τοποθετήσεις. Πολύ πιο δύσκολο είναι το έργο εκείνων που τοποθετούνται και πολύ πιο εύκολο είναι το πρόβλημα εκείνων που λένε ότι α, δεν υπάρχουν μεταβολές κλιματικές και είναι αυτή η τοποθέτησή τους. Τι γίνεται σε σχέση με την παρακμή των βιομηχανιών στην Ευρώπη και πώς μπορεί να σταματήσει και ακριβώς εδώ σε σχέση με την καινοτομία και την αηφορία δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Μόνο που κάνουμε το λάθος να μην χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες δεν δίνονται, δεν έρχονται μόνες τους, δεν πέφτουν από τον ουρανό και σωστά το είπες Chris Davis εσύ πιο πριν ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σχεδιασμού, βεβαιότητα σχεδιασμού, ότι πρέπει να αποσταλούν τα σωστά μηνύματα. Χρειάζεται η βιομηχανία αυτά τα μηνύματα. Προέρχομαι από μια χώρα όπου ελήφθη μια θεμελιωδέστατη απόφαση. Αυτή η απόφαση για την εγκατάλειψη τη πυρηνική ενέργεια είναι δεδομένη. Αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να υπάρξει βεβαιότητα και ασφάλεια σχεδιασμού χωρίς να καταργηθεί το πλαίσιο σχεδιασμού. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ένας εξαιρετικός ποταμός, όχι ορίνος, αλλά ένας μικρότερος, αλλά πολύ όμορφος ποταμός, αυτός ε, έχει ανασχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μην ε, υπάρχει εκεί ε, κάποιος πυρηνικός σταθμός. Πρέπει έτσι να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα και την επιτάχυνση της καινοτομίας που προετοιμάστηκε και σχεδιάστηκε να την υλοποιήσουμε. Μετά έχουμε και την, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω πρόεδρε, δεν έχω χρόνο έτσι, τέλειος, έληξε ο χρόνος μου. Έχουμε την επισήμαση του Chris Davis ότι στο μέλλον δεν θα έπρεπε να αποτύχει για άλλη μία φορά μία έκθεση για το περιβάλλον εννοούσε ε, τον συνάδελφο, τον οποίο εκτιμώ εγώ ιδιαίτερα και που απέτυχε η έκθεσή του και δεν εγκρίθηκε. Λοιπόν, το να έχουμε την δυνατότητα να υπάρξει ένα, μια τοποθέτηση από αυτών των θεμάτων που θα επιτύχουμε εταίρους και συνενετικά εταίρους για να μπορέσουμε να περάσουμε και να εγκριθεί αυτή η έκθεση και σε σχέση με το 20% θα πρέπει 30% να έχουμε υπόψη μας ως στόχο. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε το πράσινο εφαλτήριο με το οποίο θα προχωρήσουμε, να κάνουμε συμφωνίες μεταξύ μας για να είναι βιώσιμες και να μπορέσουν να εγκριθούν. Ευχαριστώ. Τι θα ήταν τώρα το, το συντηρητικό εφαλτήριο, μια και ανέφερε το πράσινο εφαλτήριο. Παρακαλώ εσείς. Thank Τον Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καλό το ότι συχνά το πράσινο τμήμα της συζήτησης ε, τονίζεται σε αυτά τα θέματα. Από την άλλη πλευρά όμως ε, για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς αποδυναμώνονται όσον αφορά την περαιτέρω διαδικασία στο Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων και μετά αποδυναμώνονται στο Συμβούλιο. Κάποιοι πρέπει να υποστηρίξουν την, το κοινό νου και την λογική στην προσέγγιση αυτών των πραγμάτων. Δεν είμαστε υπέρ ενό πράσινου λόμπου, ε, λόμπι, αλλά να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία. Τι μπορούμε να κερδίσουμε σε σχέση με αυτή την πορεία που ακολουθούμε. Τα στοιχεία μας λένε ότι μέχρι το, κατά το 2009 οι εκπομπές ήταν κατά 17,3% χαμηλότερες από ότι το 1990. Εννέα χρόνια απέχουμε από το 2020 σήμερα και φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο να πετύχουμε πολύ κοντά τον στόχο του 20% μείωση. Και ας, πάμε, να είμαστε, πιο φιλόδοξοι και ας υιοθετήσουμε έναν υψηλότερο στόχο μείωση θα, όπως είπε ο Νταν Γιώργενσεν, θα μπορούσαμε να έχουμε το 40%. 40% για το 2030 θα μπορούσε να είναι χαμηλός στόχος μείωσης. Ας το λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο οδικός χάρτης, να ενδυναμωθεί και τουλάχιστον να τον υποστηρίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το κόστος αναμένεται ότι θα είναι 270 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο μιλητής, ετήσια. Αν όμως υπολογίσετε τι θα, τι θα εξοικονομήσουμε όσον αφορά τις εισαγωγές ενέργειας, από 170 έως 320 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά τα ποσά. Και φυσικά το σενάριο των υψηλότερων τιμών ενέργειας είναι εκείνο το οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε η εξοικονόμηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που θα δαπανηθούν για να επιτευχθεί αυτός ο οδικός χάρτης. Θα έχουμε και 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και πέρα από την εξοικονόμηση όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα θα έχουμε επιπλέον και 17 δις ευρώ ετήσια το 2030 και 38 δις ευρώ ετήσια το 2050 κέρδους που θα σημειωθεί από την βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα που θα πετύχουμε. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι φυσικά να αυξήσουμε τις επενδύσεις και αυτή η αύξηση κατά 1,5% που αναμένεται να οδηγήσει σε μια αναλογία προς το ΑΕΠ θα είναι κατά 20,5% μικρότερο σε σχέση με αυτά τα οποία επιτυγχάνει η Ινδία ή η Κορέα. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι επιτακτική ανάγκη αν δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω σε σχέση με άλλες χώρες και για να πετύχουμε δεσμευτικούς στόχους και αν δεν θέλουμε να μετεγκατασταθούν οι βιομηχανίες μας σε άλλες χώρες αλλά να παραμείνουν στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε Κρήτον. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και τώρα μπορεί ίσως να είναι μια πρόκληση πνευματικά ή διανοητικά, πολιτικά να σκέφτεται κανείς ένα χρόνο πλαίσιο 40 ετών, αλλά όμως όλα αυτά θα πρέπει σε σωστές διαστάσεις να τα δούμε και στο σωστό πλαίσιο να τα εντάξουμε. Δεν είναι μόνο εδώ το θέμα του να υπάρξει κάποιο ερώτημα για το αν υπάρχουν κλιματικές αλλαγές ή όχι, ή να αρνηθεί κανείς αυτές τις αλλαγές, αλλά να δούμε ποιους στόχους θα θέσουμε και πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε σωστούς στόχους και τι θα κάνουμε αν υιοθετήσουμε την προσέγγιση ότι θα υπάρξουν αυτές οι αλλαγές και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Εδώ, σε σχέση με την αξιοπιστία της ανθρώπινης προόδου, δεν πρέπει να τα δούμε μηχανιστικά τα πράγματα σε ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο, διότι το αργότερο από την κβαντική φυσική γνωρίζουμε την απροσδιοριστία, την αρχή της απροσδιοριστίας και ότι δεν είναι δυνατόν να όλα να προ δικαστούν ακόμα και σε σχέση με την θεωρία της σχετικότητας ε, του Άινστάιν ε, δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να προδικάσουμε το τι ε, είναι δυνατό να συμβεί. Με την κβαντική μηχανική και φυσική αποδείχτηκε αυτή η απροσδιοριστία. Τώρα πρέπει στο πολιτικό επίπεδο να δράσουμε και να εντάξουμε τα πράγματα στα σωστά τους μεγέθη και είναι ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς τι θα συνέβαινε αν στην υποθετική εκείνη περίπτωση που αλλά ας σκεφτούμε ποιος θα σκεφτόταν τη δεκαετία του 80 ή τη δεκαετία του 70 ότι κάποτε θα κατέρεε το σίδηρο, το σίδηρο παραπέτασμα και η Σοβιετική Ένωση ήταν ασύλληπτα πράγματα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και να προδικάσει τις εξέλιξεις στο μέλλον. Και για αυτή την τεχνολογική επανάσταση, εσύ ο ίδιος ε, πρόεδρε ανέφερε σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα επιβάλλει κανείς ε, ε, και ούτε και είναι δυνατόν με την θεωρία της σχετικότητας να επιβάλλει κανείς κάποια πράγματα. Κανείς δεν προέβλεψε την εποχή του διαδικτύου και της επανάστασης της πληροφορικής με την ανάπτυξη των σωστών ε, συνθήκων πλαισίου πλαισίου έγιναν δυνατά και εφικτά αυτά, αλλά πρέπει κάπως να είμαστε πιο ταπεινόφρονες και να σκεφτούμε τι είναι πραγματικά δυνατόν να πετύχουμε και τι δεν μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά που μπορούμε να πετύχουμε και αυτό πρέπει να αναφέρει το έγγραφο είναι η απεικόνηση της ε, σωστής της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Και πρέπει λογικά να είμαστε συνεπείς, να υπενθυμίσω ότι η μόνη Ήπειρος, αν θέλετε, σε παγκόσμια κλίμακα όπου οι τιμές ε, για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του, του, ε, του άνθρακα έχουν εισαχθεί και λειτουργούν δεν χρειάζεται να, να φοβόμαστε ότι άλλες ε, χώρες ε, θα, εφόσον εμείς είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το επίπεδο στο παρελθόν, θα μας αφήσουν πίσω και θα μείνουμε ουραγοί. Λοιπόν, ή το χρειαζόμαστε σε σχέση με τη διατήρηση της ε, τεχνολογικής μας, ας το πω έτσι, διαφοράς που μας χωρίζει από τις άλλες χώρες είτε δεν τα χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε όλα αυτά, να δούμε αν είναι αναγκαία. Και σε αυτή τη γραμμική τεχνολογική πρόοδο μέχρι το 2005 το να προβλέψουμε και να καταδικάσουμε κάποια πράγματα όπως ε, αναφέρεται ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα περισσότερα από αυτά που έχουν σχεδιαστεί, όλα αυτά ακούγονται, ας το πω έτσι, τουλάχιστον αβάσιμα ή όχι τόσο πιστικά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ε, χάσουμε την επαφή στην πραγματικότητα που είναι αναγκαίος μύτος της Αριάδνης ε, για την ανάπτυξη των θέσεών μας. Θα πρέπει μια δεσμευτική απόφαση να ληφθεί μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ρίχαρτ Ζέιμπερ. Εδώ θα έπρεπε ανεκδοτολογικά να αναφέρω κάτι. Προειδοποιήθηκε και δόθηκε προειδοποίηση να μην ε, κάνουμε προγνωστικά για μία περίοδο 40 ετών για την έκθεση για την βιοπικιλότητα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Βερολίνο ε, είχαμε τον χαιρετισμό και σε σχέση με αυτά τους δεινοσαύρους, τεράστια ζώα που έζησαν πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια. Ο Μεσαίος βρίσκεται πιο κοντά σε μάσα από ότι στους μεγάλους ε, δεινοσαύρους και έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια ο Μεσαίος αυτός δεινόσαυρος στο μέγεθος και σε σχέση με την ε, περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης 200 ετών κάψαμε όλα τα ορυκτά καύσιμα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε όλη αυτή την τεράστια περίοδο. Ας μην μου πει κανείς ότι αυτό δεν έχει επιπτώσεις για τον πλανήτη. Αυτά τα 40 χρόνια είναι ένα μηδαμινό στοιχείο σε σχέση με την ιστορία της γης και το ίδιο το μυαλό μας, η φαιά μας ουσία δεν είναι σε θέση αυτά τα σύλληπτα πράγματα να τα συλλάβει. Γι' αυτό το σενάριο του 2050 ως πρόγνωση είναι το ελάχιστο που πρέπει να σχεδιάσουμε και να προβλέψουμε και αν πούμε ότι δεν έχει ούτω ή άλλω ο άνθρωπο καμιά επιρροή στι αλλαγέ του περιβάλλοντο, ε, τότε δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και θα πάνε όλα του κάκου. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείω από το χρονικό πλαίσιο. Άννα Χόσπαχ, και εδώ θα πρέπει να επιμείνω τρία λεπτά η κάθε παρέμβαση. Παρακαλώ, Άννα. Er ναι, Πρόεδρε, δεν είναι βέβαια δίκαιο να περιορίσετε το δικό μου χρόνο ομιλία. Θα προσπαθήσω όμω να κάνω ό,τι μπορώ. Όπω έχουμε τώρα τα πράγματα, είναι μεγάλες διαφορέ που εμφανίζονται στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030 μπορεί να φαίνεται πολύ μακριά, αλλά τα οράματα για το μέλλον φαίνεται ότι ορισμένα κράτη-μέλη τα θεωρούν πολύ δύσκολο να σεβαστούν, να τα λάβουν υπόψη τους. Και όμως είναι, οι χώρες, είναι πολλές οι χώρες οι οποίες έχουν, ε, α, κηρύξει, έχουν ανακηρύξει νέες πολιτικές. Θέλουμε 40% νέων πηγών ενέργειας ε, στα επόμενα 9 χρόνια και νομίζω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Όμως έχω την εξή δυσκολία. Εάν δεν λαμβάνουμε σωστά ε, μέτρα, δεν μπορούμε καν να επιτρέψουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή της έρευνα στους νέους τεχνολογικούς τομείς. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πολλά. Δεν χρειάζεται να καταγράφουμε διεξοδικούς καταλόγους ε, του τι πρέπει να γίνει. Σε ορισμένε περιπτώσει είναι πιο εύκολο να περιορίσουμε τις, να εστιάσουμε δηλαδή τα μέσα μας και την προσοχή μας σε ε, έρευνα σε, ορισμένες, ε, σε ενέργεια τομείς ενέργειας που ήδη υπάρχουν και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, όπως είναι η υδροηλεκτρική, όπως είναι η ηλιακή, η αιωλική ενέργεια που έχουμε και στη Δανία και πρέπει να κοιτάξουμε και την ενέργεια που παράγεται από τα απόβλητα. Και μίλησα μόνο για δύο λεπτά, Πρόεδρε. Μπράβο σας, μπράβο σας, λέει ο Μέσα δύο λεπτά, συγχαρητήρια. Ανδρέα Τζαρόνι, επόμενος μιλητής. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κρυς Ντέιβις για το έγγραφό του. Το οποίο συμμερίζομαι απόλυτα. Ο συνάδελφος μας καλεί να κάνουμε μία επιλογή. Από ποια μεριά θέλουμε να σταθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει μία αξιόπιστη απάντηση για την, για την αύξηση της θερμοκρασίας και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει αρχηγικό ρόλο σε αυτό το μέτωπο. Χρειάζεται να υπάρξει ένα δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ των βιομηχανοποιημένων χωρών. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρνούνται το φαινόμενο παρά τα, τα, τα, εμφανή αποτελέσματα όπως είναι το λιώσιμο των πάγων στην Ακτική τις προάλλες δύσπιστος άκουσε έναν συνάδελφο να τοποθετείται λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης της γης. Και σήμερα άκουσα περίεργα πράγματα από κάποιον. Νομίζω ότι αν κάποιος συνεχίζει να το τραβάει προς αυτήν την κατεύθυνση θα ξεπεραστεί και τεχνολογικά από τις τρίτες χώρες, κυρίως στον τομέα των εναλλακτικών ενεργειών και της ηλιακής ενέργειας. Θα υπάρξουν επιπτώσεις στη γεωργία και σε παγκόσμιο επίπεδο διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη βιοποικιλότητα πολλά αποδημητικά πουλιά υποφέρουν σήμερα από τις κλιματικές αλλαγές, υπάρχουν και άγρια ζώα τα οποία έχουν αλλάξει συμπεριφορές, χρήσιμα έντομα επίσης υποφέρουν. Σε πολλές χώρες βλέπουμε τα φύκια να πολλαπλασιάζονται κυρίως στις ακτές όπως επίσης και σε παραθεριστικούς ε, παραλιακούς ε, τόπους ε, μπορούν να προκύψουν νέες ασθένειες, οι άνθρωποι μπορούν να, έχουν, να, να, να, αρρωσταίνουν με περίεργες αρρώστιες οι οποίες δεν υπήρχαν ποτέ σε ορισμένες περιοχές. Χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ακούσαμε τον Διευθυντή του Κέντρου για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών, τον κύριο Σπρέγκερ, ο οποίος είπε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη διάδοση των ασθενειών. Αυτή η έκθεση για το φύλλο πορείας για τη μετάβαση στην ε, για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050 αποτελεί ένα καταπληκτικό μέσο για να πιέσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να προχωρήσουμε γρήγορα και να αποφασίσουμε νωρίς. Πρέπει να ληφθεί μια σαφής απόφαση και να πιστεί όλο το Κοινοβούλιο για μία από τις πιο σημαντικές, όπως λέχθηκε, ψηφοφορίες της κοινοβουλευτικής μας θητεία. Πρόκειται για μία ισορροπημένη και φιλόδοξη έκθεση. Ευχαριστώ κύριο Λίσσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και, και, παρότι δεν έχουμε χρόνο, μια και έχει γίνει όλη αυτή η συζήτηση που έγινε, θέλω να κάνω μια συζήτηση επί της ουσίας. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να παραπέμπουμε στη θέση στέρα όταν μιλούμε για, την, ε, για τον σχετισμό μεταξύ ε, οικονομίας και κλιματικών αλλαγών, γιατί η οικονομική κρίση του 2009 είχε, νομίζω, προβλεφθεί ως ε, το λιγότερο κακό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Ένας από τους ηγετικούς οικονομολόγους, ηγετικές προσωπικότητες της οικονομίας στον κόσμο, ο κύριος Στέρν είχε προβλέψει ότι εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές αλλαγές δεν θα μπορέσουμε να ανθέξουμε οικονομικά τις εξελίξεις. Πολλές λοιπόν ε, οι αντιδράσεις σε αυτό, αλλά ερευνητής στα θέματα του, τα κλιματολογικά προσπαθούσε να με πείσει <clears throat> και για την οικονομική διάσταση της υπόθεσης αυτής προσπαθούσε να, να μου πει λοιπόν να ε, μου, με βάλει να αναζητήσω οποιαδήποτε ιατρική περίπτωση, κρούσμα, φάρμακο, αγωγή, διαδικασία που να απασχολεί τόσους πολλούς ιατρούς στον κόσμο για να κάνει την αντιπαραβολή με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που απασχολεί όλους τους ε, επιστήμονες στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ε, ως γιατρός στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, εάν δω ότι και εγώ και άλλοι 3.000 συμφωνούν στην ίδια, αγωγή, στην ίδια διάγνωση και στην ίδια αγωγή, προφανώ και πρέπει να εφαρμόζω την αγωγή. Αυτή είναι λοιπόν, αυτό είναι ο κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή. Είναι φιλόδοξη, ίσω είναι υπερβολικά φιλόδοξη η επιλογή τη, Είναι ένα καλό δρόμο, μιλούμε για μακροπρόθεσμου στόχου. Ταυτόχρονα όμω, μιλούμε και ε, υπάρχει ανάγκη και για πιο συγκεκριμένε πρωτοβουλίες. Βεβαίως και η γραμμική προσέγγιση από το 90 στο 2050 είναι πολύ πιο μεγάλη πρόκληση από αυτό που συζητούμε τώρα, αλλά έχουμε ξεκινήσει μια προσέγγιση η οποία θα μας πάει σε αυτό το ορίζοντα 50 ετίας, 50 ετίας, με στάδια. Έχουμε ξεκινήσει από το 2005, έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε αν η γραμμή έχει τραβηχθεί σωστά, εάν τα στοιχεία που ακολουθούμε είναι ευσταθούν και αν οι επιλογές μας είναι σωστές κάθε τόσο. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν στη χρήση ενέργεια είναι αλληλένδετη φυσικά με αυτόν τον οδικό χάρτη και έχουμε το στόχο του 2020 που θα πρέπει να τηρηθεί. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να προσδιορίσουμε και στόχου ε, συνεπείς, συμβατούς με τον περιορισμό του δεξιού του άνθρακα για το 2030-40-50 και να υπολογίσουμε ότι μπορεί να μην χρειάζεται νέο ηλεκτρικό ρεύμα και άρα δεν χρειάζονται νέες, ε, νέα δίκτυα και νέο, νέες ικανότητες. Καλή λοιπόν η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η προσπάθεια να γίνει πιο συγκεκριμένη και νομίζω δεν πρέπει να την επικρίνουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω στις βασικές αρχές που έχει οθετήσει αυτή η στρατηγική. Ευχαριστώ κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα και για να μην υπησέτω στην ουσία πρέπει να πω ότι αναπτύχθηκαν τέλεια από τους συναδέλφους μου τα επιμέρους στοιχεία, αλλά απλά ήθελα να πω ότι σε σχέση με την ε, ε, ισπανική παρέμβαση, αλλά το τελευταίο σημείο όπου κάνει λόγο ο κύριος Κρίς Ντέιβις για τη δική μας ευκαιρία που μας προσφέρεται, δύο μικρές παράγραφοι εμφανίζονται που διαβάζω τη μία λέξη προς λέξη. Σε περίοδο πολέμου τα πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα. Βρίσκονται χρήματα, μειώνεται η γραφειοκρατία, λαμβάνονται αποφάσεις. Και έχω την εντύπωση, εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου. Κατανοώ βέβαια αυτό που θέλει να πει ο κύριος Κρίς Ντέιβις ε, ρητορικά σε σχέση με αυτή την περίοδο περίπτωση καταστροφής, την περίπτωση πολέμου, για να μας δείξει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, αλλά θα παρακαλούσα τον κύριο Ντέβις <laughs> και όποιον είναι αρμόδιος να μην έχουμε τέτοιες γραμμές, τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί α, διαβάζοντας αυτή την παρέμβαση μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ο καλύτερος όλων των δυνατών κόσμων είναι εκείνος στον οποίο υπάρχει πόλεμος ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Κρις Ντέιβις για την αμεσότητα της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν έχουμε εμπόλεμη περίπτωση, δεν είναι περίπτωση πολέμου, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό και έχει τεράστια σημασία και πρέπει οπωσδήποτε και οπωσδήποτε συμμερίζομαι του ότι να λυθούν αποφάσεις για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ωστόσο όμως με κανένα τρόπο δεν μας δικαιολογεί αυτό το να είμαστε υπέρ μιας περίπτωσης ε, πολέμου ή εμπόλεμης κατάστασης. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί με αυτά τα πράγματα εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σοφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα όμως να πω ότι το έγγραφο του κυρίου Ντέιβις είναι ένα πολύ καλό έγγραφο και άκουσα και το ανέκδοτό σας και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τη μείωση της ρήπανσης και να συμμετέχουμε σε αυτό. Όμως Πιστεύω ότι πέρα από αυτή την ιδέα του να καταναγκάσουμε ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις μας με νέους κανόνες και δεσμεύσεις που τις επιβάλλουμε όταν αντιμετωπίσουν, θέλουν να παράγουν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να ορίσει μία νέα ωραία βιομηχανική πολιτική ανταγωνιστική που να τίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, που να πηγαίνει προς την έρευνα, να εφαρμοστεί μία ε, φιλόδοξη ε, ε, πολιτική έρευνας, μέσα από τις πολιτικές μας, την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχή, έχουμε τα μέσα για να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία φαίνεται ότι τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ της περιφερειακής πολιτικής με ένα κεφάλαιο έρευνα και καινοτομία δεν καταναλώνεται ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δεν... Ορισμένα κράτη απορροφούν λιγότερο από το 20% ενώ βρισκόμαστε και ενώ είμαστε δηλαδή σε ένα επταετές ε, πρόγραμμα στα δύο τρίτα του, του, του προγράμματος. Χρειάζεται φιλόδοξη πολιτική για το περιβάλλον. Φυσικά και συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει αυτό να το κάνουμε σύμβατα με μια πολιτική έρευνας και βιομηχανίας φιλόδοξες ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα ενέργεια για, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε ας πούμε αέριο, από σχιστολιθικό αέριο, χρειάζεται να έχουμε και την απαραίτητη τεχνολογία να μπορούμε να το παράγουμε χωρίς να ρηπαίνουμε. Προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Αυτά ήταν ε, τα στοιχεία της συζήτησής μας πολύ πλούσια και από πλευράς παρατηρήσεων και τοποθετήσεων αξίζει να συζητήσουμε μέσα σε ένα τέτοιο πλούσιο πλαίσιο. Θα λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος από την Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστούμε τον κύριο Ντέιβις. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή του, το έγγραφο βάσεως. Πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση, πολύ ζωντανή. Κάποιες παρατηρήσεις χωρίς να επισέλθω σε πολλές ε, λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που ε, προέκυψαν στη συζήτηση. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση και σχετική με το συσχετισμό ε, ως προς το διεθνή μας προγραμματισμό. Είμαστε μόλις μερικούς μήνες πριν από τον Τουρμπάν. Ωστόσο πρέπει να ξέρουμε ότι και στο Κανκούν οι ηγέτες των κρατών του κόσμου συμφώνησαν στην αύξηση των δύο βαθμών με βάση και τα στοιχεία του IPCC και άρα είναι ένας δεκτός από τις χώρες όλου του κόσμου, τους ηγέτες όλου του κόσμου στόχος αυτός πλέον. Στο Κανκούν και οι αναδυόμενες και οι ανεπτυσσόμενες ε, οικονομίες έκαναν ε, προτάσεις σχετικές ε, με το 18% στις παγκόσμιες εκπομπές. Άρα έχουμε δεσμεύσεις πλέον σε ολόκληρο το κόσμο. Και παραλαμβάνω, δεν αρκεί να είναι βέβαια να είμαστε συμβατοί με το στόχου των δύο ε, βαθμών, αλλά τουλάχιστον αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα κάποια σχόλια ως προς τη φύση αυτού του οδικού χάρτη. Έγινε λόγος ε, για το αν θα είναι ένα σχέδιο, μία πρόβλεψη για το πώς κόσμο κόσμος θα διαμορφωθεί το 2050. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό με τον οδικό αυτό χάρτη να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να διδαχθούμε από το τι μπορούμε να κάνουμε με βάση την προηγούμενη μας εμπειρία και για τα επόμενα βήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να επενδύσουμε, ποιες είναι οι ε, τεχνολογίες, οι κέρυες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση, που πρεπει να επενδυσουμε ποιε ειναι οι τεχνολογιες οι κερυες στις οποιες θα πρεπει να δωσουμε περισσοτερη εμφαση που μπορει να βρει η Ευρώπη καλύτερες ευκαιρίες, που θα πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίες και από την άλλη κάποιες, επί τη βάση αυτής της, ε, αυτών των γνώσεων, αυτής της αντίληψης, αυτής της νοοτροπίας, να προχωρήσουμε σε πολιτικές επιλογές. Ορόσημα. Τα ορόσημα αποτελούν βεβαίως κρίσιμη σημασία στοιχείο αυτού του οδικού χάρτη. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζητεί και ο κλάδος. Περισσότερη δηλαδή σαφήνεια, ε, διάβγεια για το μέλλον, για να μπορούν να ευθυγραμμιστούν στόχους. Έχει υποθεί και στο παρελθόν ότι πρέπει να έχουμε στόχους που θα μας ε, πάνε για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια. Και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία. Στόχοι βέβαια δεν είναι αυτή, είναι απλώς ορόσημα γιατί στόχοι όπως στόχοι του 2020 συνεπάγονται και πιστώσεις ε, διεθνείς, σε διεθνές επίπεδο με τις εκπομπές και τη μείωση των εκπομπών. Και επίσης ετέθη ένα ζήτημα σχετικό με την γραμμικότητα. Γραμμική δεν είναι η πρόταση και υπάρχει σαφή λόγο, διότι ανταγωνιστικέ θα γίνουν ορισμένε από τι τεχνολογίε αυτέ μόνο αργότερα. Είτε πρόκειται για, τις, ε, για την χρήση περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στι μεταφορέ ε, ή άλλε επιλογέ. Μόνο μετά το 2025 μπορούμε να έχουμε πρακτική χρήση του. Επίσης, το κόστος για τον καταναλωτή που ερώτησε κάποιος ομιλητής είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό, όπου θα πρέπει πιστεύω να γίνει μια ανάλυση περαιτέρω ε, του κόστους ανοικοκυριό σύν το χρόνο, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια πρώτη ιδέα ως προς τις επενδύσεις που θα χρειαστούν και την εξοικονόμηση σε ορυκτά καύσιμα ε, χάρη στις επενδύσεις αυτές. Επενδύσεις που υπολογίζουμε στα 270 δισεκατομμύρια το χρόνο κατά μέσο όρο, και αντίστοιχη εξοικονόμηση καυσίμου, πολύ σημαντικό στοιχείο δηλαδή, αλλά επίσης αυτό συνεπάγεται και μεγάλη μετακύληση της χρονικής στιγμής, ε, μάλλον μεγάλη ναι, μετακύληση του βάρους και της χρονικής στιγμής στην οποία θα γίνει αυτή η επένδυση. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να προκαταβάλουμε τρόπον την άτσι σε αυτές, στο κόστος αυτό. Επίσης, ακολουθούμε τις πολιτικές ε, για την πυρηνική ενέργεια που έχουν τα κράτη-μέλη επιλέξει με αυτό το δεδομένα κάνουμε του τους υπολογισμού μας, αυτά φυσικά πριν από τη Φουκοσίμα. Στη Γερμανία υπήρχε ήδη η πρόβλεψη να καταρριφθεί η πυρηνική ενέργεια και μετά βέβαια άλλε αποφάσει. Πάντω στο δικό μα το σενάριο για το 2050, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον δεν βλέπουμε πυρηνικά στη Γερμανία, δεν την υπολογίζουμε πυρηνικά στη Γερμανία. Αλλά όπω είπα, βασιζόμαστε στι επιλογέ που έχουν ήδη κάνει τα κράτη-μέλη για τα πυρηνικά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας, εξηγήσεις εκ Επιτροπής. Θέλει ο Chris Davis να κλείσει τη συζήτηση με τις παρατηρήσεις του. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίλο, που ήταν ο συντάξης για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα υπενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι έχουμε την ε, διάταξη του άρθρου 50 του κανονισμού. Η αρμοδιότητα τη της Επιτροπής μας έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές και τα δίκτυα. Ως εκ τούτου, οι αδίποτε ε, τροπολογίες στα θέματα αυτά πάνε στον κύριο Πυρίλο και την έκθεσή του με προθεσμία για κατάσταση τροπολογιών την επόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος κύριε Πυρίλο, έτσι δεν είναι, Του πω την επόμενη εβδομάδα. Για τη δική μου έκθεση πάμε για μετάφραση κάπου στα τέλη του μήνα και ε, προβλέπω συνάντηση με τους ε, σκιώδεις σε δύο-τρεις εβδομάδες, πριν δηλαδή από τη μετάφραση, για να προλάβουν να σωματώσω κάποια σχόλια. Κάποιες προτάσεις που ακούστηκαν με ενδιαφέρουν πολύ, θα ήθελα να τις ε, συζητήσω για τον κύριο Ρώση, Φερρυπίν, για τον κύριο Κράμερ. Είναι πολλά αυτά που είπαν. Και ο κύριος Γιώργενσεν όμως νομίζω τα, ε, τις κάλυψε τις θέσεις αυτές ικανοποιητικά και άλλωστε εν γέννη νομίζω ακούστηκαν ε, επιχειρήματα που ε, αποδεικνύουν ότι ορισμένε θέσει ήταν ασφαλμένε. Δεν θέλω λοιπόν να επισέλθω στις λεπτομέρειες. Αλλά για την έκκληση του Καρλ Χάιντ να υπάρξει μια εταιρική, συνεταιρική στάση εδώ. Ναι, προφανώς και θα ήταν καλό να μπορούσαμε να έχουμε συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να γίνει με καλά αποτελέσματα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια σε προτάσεις που ελπίζω θα στηρίξουν ε, τον οδικό χάρτη και θα τον ε, προαγάγουν περισσότερο. Βεβαίω και θα ήταν καλό να έχουμε συνένεση ως προς, ε, προς τα ορόσημα. Ελπίζω επί την άλλη να μην ενόχλησα πολλούς συναδέλφους με την πολύ απερίφραστη διατύπωση που ακολουθώ μερικέ φορέ. Ξέρουμε ότι οι πόλεμοι πολλέ φορέ οδηγούν σε νέε προκλήσει και επιτυχίε, επαναστάσει. Ναι, αλλά και οι νέοι στόχοι επίση, όπω ε, η επιλογή των Αμερικανών στη δεκαετία του 60 να φτάσουν μέχρι το φεγγάρι στη δεκαετία του 60, δίνει νέε δράσει, δίνει νέους, ε, νέο κέρδο, νέα επιτυχία. Επομένως υπάρχει λόγος να στηρίζουμε νέους ε, στόχου. Το 2050 μπορεί να μα φαίνεται πολύ μακριά και μάλλον θα είμαστε ορισμένοι σε ένα ξύλινο, περισσότεροι μάλλον εξημών, σε ένα ξύλινο κουτί να ε, προσφέρουμε λίπασμα στα ραδίκια. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία αυτού του στόχου και το 2040 είναι πολύ σημαντικός στόχος ε, και ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, κοιτάξει το θέμα αυτό και από την έποψη της ενέργειας μέσω της Γενικής Διευθύνσης Ενέργειας για να εξετάσει εάν μπορεί είτε να μείνει στην, ε, στο στόχο του 2050 είτε να ορίσει ορόσημα. Η εταιρική σχέση που αναφέρθηκε ο Καλ Χάιντ. συνεπάγεται ότι ορισμένοι εξημών εδώ θέλουν ε, ε, φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό των ε, αερίων του θερμοκηπίου, να συμβάλλουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αυτόν στην βελτίωση του, της κατάστασης τον κόσμο, αλλά και να βοηθήσουν ταυτόχρονα και τις επενδύσεις και τα κεφάλαια. Πολλοί είναι αυτοί από τον κλάδο και κυρίως από την ενεργειακή παραγωγή που μας ζητούν ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή σαφή μηνύματα και επαρκή ε, ασφάλεια δικαίου ώστε να μπορούν ε, να ε, προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις που συνεπάγονται εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό νομίζω πρέπει να πράξουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας και επί τη βάση των συζητήσεών μας θα ετοιμαστεί φαντάζομαι και το σχέδιο της εκθέσεως. στην συνέχεια την ξέρετε πώ πάει η διαδικασία. Ευχαριστώ, Chris που ανέλαβε στην πορεία μέχρι το σχέδιο εκθέσεως. Και τώρα περνάμε στο σημείο 15. Άλλο ένα χάρτη πορεία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών με συντάκτη τον κύριο Μπόγκουσλαφ Σόνικ για γνωμοδότηση. Επί της ουσίας αρμόδια η Επιτροπή των Μεταφορών με τον κύριο Ματσίου Γκρούς. Έχει λόγο, Μπογουσλάφα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τις μεταφορές. Οι μεταφορές είναι τα θεμέλια της οικονομίας μας, της κοινωνίας μας και συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων θέσεων απασχόλησης. Η ανάπτυξη των μεταφορών, λοιπόν, πρέπει να είναι αηφόρου χαρακτήρα, με αηφορία. Είναι ένας παγκοσμιοποιημένος ε, ο οικουμενικός τομέας. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και πολλές πρωτοβουλίες χρειάζονται στα πιο διαφορετικά επίπεδα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, στη γνωμοδότησή μου, επισημαίνω ότι όπου είναι δυνατόν πρέπει να υπάρχει μια μετάθεση, μετάθεση προς μη εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων στα οχήματα με κινητήρες, διότι δεν θα είναι Αυτά τα οχήματα που δεν θα χρησιμοποιούν τέτοια καύσιμα δεν θα είναι επιβαρυντικά στο περιβάλλον και στο κλίμα με τις εκπομπές τους. Πρέπει λοιπόν να μην και με ορυκτά καύσιμα. Δεύτερον, οι εκπομπές ρήπων σε σχέση με την ενέργεια θα πρέπει να μειωθούν με την χρήση νέων τεχνολογιών στην μηχανές καύσεως. Υποστηρίζω έρευνα σε τέτοιες καινοτόμες τεχνολογίες και τέτοια τεχνολογία για τις μεταφορές. Μαζική μετάθεση απαιτεί χρόνο. Γι' αυτό οι δράσεις που θα γίνουν μέσα σε αυτές τις διεργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια την πραγματικότητα επιτόπου, στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προάξει, να προαγάγει και να υποστηρίξει οικονομικά πανευρωπαϊκή δίκτυα, κοινοτικά πανευρωπαϊκά δίκτυα σιδηροδρόμων ώστε να μπορέσουν να περάσουν τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αγαθών στις σιδηροδρομικές μεταφορές και να μεταφέρονται αυτά τα φορτηγά με σιδηροδρόμους. Η σύσταση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εκείνες τις περιφέρειες και περιοχές όπου υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς αυτό. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε τις μελλοντικέ μας δράσεις λοιπόν σε αυτό το επίκεντρο να μειωθούν οι διαφορές σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών όσον αφορά διαφορετικές περιφέρειες και περιοχές κρατών μελών. Έχω συνειδητοποιήσει ότι οι νέες τεχνολογίες όσον αφορά τις μεταφορές είναι και χρονοβόρες και χρηματοβόρες Γι' αυτό η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και ο περιορισμός τους είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων στις μεταφορές συνολικά. Θα ήθελα να τονίσω επίσης την σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιου είδους δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδια θα έπρεπε να ξεκινήσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τέτοιες εκστρατείες υπέρ νέων εναλλακτικών δυνατοτήτων και τύπων και ε, τρόπων μεταφορών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόνικ. Έχουμε σκιώδη εισηγητή, την Ινέσα Αγιάλα Σέντερ. Παρακαλώ Ινέσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σόνικ για το ότι κατάφερε σε τόσο λίγες παραγράφους να συμπυκνώσει όλη αυτή τη σημαντική συζήτηση που είδαμε και προηγουμένως δηλαδή ε, πρόκειται για συζήτηση όπως το θέτει η Κομισιόν εν ώψη του, της περίοδου μέχρι το 2050 για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σε τομείς κυρίως που χρειάζονται μεγάλες περιόδους μπροστά τους ε, για να προσαρμοστούν και να αλλάξουν αλλαγή των υποδομών, αλλαγή των οχημάτων, αλλαγή των καψίμων ε, αλλά κυρίως και βασικά προβλήματα σχεδιασμού. Ακόμη και το θέμα της ε, ε, πολεοδομίας, οι πόλεις μεγαλώνουν και απαιτούν ε, υποστήριξη από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιασμού για να μπορέσουν να αλλάξουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος το σημαντικό είναι να μην μειώσουμε την κινητικότητα. Πρόκειται για μια ρηψοκίνδυνη επιλογή. Αλλάζει έναντι του παρελθόντος. Στο παρελθόν είχαμε ένα πρόβλημα χάσματος μεταξύ κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. και δεν υπήρχε οικονομική ανάπτυξη αν δεν είχαμε κινητικότητα. Δεν μπορούμε εμείς να μειώσουμε την κινητικότητα μόνο για να μειώσουμε. Θα... Πρέπει σίγουρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην κινητικότητα, αλλά όχι περικοπές θα ήθελα να, δει, να, εξετάσουμε βαθύτερα όλη την πολεοδομική πλευρά του πράγματος ε, την, τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, να επιμείνουμε στις συλλογικές δημόσιες υπηρεσίες, ε, τους ποδηλατοδρόμους, τα πεζοδρόμια, δηλαδή ότι έχει σχέση με ποδηλασία και πεζοπορία θα πρέπει να δούμε επίσης ε, και το λογισμικό πρόβλημα για την μεταφορά των εμπορευμάτων, ε, πώς ε, θα αντιμετωπιστεί αυτό περιβαλλοντολογικά. Διότι ναι μεν εμείς λύνουμε το πρόβλημα των μεταφορών των προσώπων αλλά τις, τα εμπορεύματα δεν τα εξετάζουμε ποτέ. Καλό θα ήταν να, δώσουμε, να εξετάσουμε και αυτό το θέμα σε αυτή τη φάση που πρέπει να δοθούν λύσεις και χρειάζονται καινοτομίε στον τομέα μεταφοράς των εμπορευμάτων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πραγματικά εκραγεί, έχει υπερπολαπλασιαστεί. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την πτυχή του θέματος. Ε, για το διεθνές ε, τμήμα, το θέμα της παγκοσμίου κινητικότητας, μεταφορές στο πλαίσιο του 2050 πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι αποφάσεις για την αεροπορία ή την αυσιπλοεία είναι από, για νέα καύσιμα, μείωση εκπομπών, ε, είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν μια τεράστια διεθνή συνιστόσα και σχετίζονται άμεσα και με το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν ε, ε, ταλαντεύσεις ε, κυρίως όταν πρέπει να ανταγωνιστούμε τις Ηνωμένε Πολιτείε κατά τη διαπραγμάτευση των διεθνών συμφωνιών θα πρέπει να θέτουμε στους ναι, θα πρέπει συγγνώμη, να μελετήσουμε το με ποιες θέσεις θα πηγαίνουμε σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Στις 19 Οκτωβρίου η Κομισιόν θα υποβάλει την πρότασή της για τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχει μια νέα διατύπωση, μια νέα άποψη και οπτική. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και εμείς την γνωμοδότησή μας για το περιβάλλον για τις αλλαγές τρόπου μεταφοράς, ε, τους σιδηροδρόμους, τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους, να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, να δούμε και το πρόβλημα της κρίσης θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος όπου θα έχουμε ε, μη καταστροφή θέσεων απασχόλησης ε, θα έχουμε ίσως και κατάργηση ορισμένων κλάδων που πιστεύαμε ότι θα ίσχυαν για πάντα. Ζητάμε λοιπόν από την Κομισιόν να εργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την διερεύνηση των πρασίνων επαγγελμάτων την ε, διαπίστωση τους, ε, την διαπίστωση νέων επαγγελμάτων και νέων ειδικοτήτων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νέες αγορές. Ε, το, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να λύσει πολλά πράγματα. Αλλά αυτά τα αυτοκίνητα βγαίνουν στην αγορά. Τι γίνεται όμως με το θέμα της ασφάλειας ή τι γίνεται με τα συνεργεία που θα πρέπει να επισκευάζουν αυτά τα αυτοκίνητα και που δεν έχουμε εμείς προβλέψει την κατάρτιση αυτών των νέων επαγγελμάτων για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές. Μετά υπάρχουν οι οικονομικές πλευρές, και το εξωτερικό κόστος. Όλα αυτά είναι πλευρές που θα πρέπει να διαπιστώσουμε και να βρούμε κίνητρα. Όχι μόνο να τιμωρούμε, αλλά να δίνουμε και κίνητρα. Εμείς έχουμε μια Ευρώπη που μεγαλώνει, όσο, που μεγαλώνει συνεχώς. Και όταν έχουμε εμεί τα εξωτερικά μας σύνορα γείτονες οι οποίοι είναι πιο δυνατοί από μας, θα πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε ορισμένες λογικές κέντρου περιφέρειας. Επίσης κύριε Σόνικ, θα ήθελα να λάβετε υπόψη και τις τεράστιες αλλαγές μεταξύ περιφερειών και κρατών στα δίκτυα ε, μεταφορών, στα δίκτυα κινητικότητες, οι διαφορές δηλαδή μεταξύ σιδηροδρόμων, ε, ε, θαλασσίων μεταφορών, αερομεταφορών κλπ. θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαφορές κινήτρων και ενισχύσεων στα διάφορα κράτη-μέλη, τα οποία το καθένα προσπαθεί να προωθήσει τα δικά του, του μέτρα, ε, μέσα συγγνώμη, μεταφοράς με το δικό του τρόπο. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θα προωθήσουμε τα πράσινα επαγγέλματα για να ενισχύσουμε αυτή τη νέα οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκυλμπράντε και μπορεί να μου πείτε ότι δεν είναι δίκαιο αλλά θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Πρόεδρε ευχαριστώ. και θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω, να είμαι στο δυνατόν πιο οικονομικός. Θα μιλήσω εκ μέρου και του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος ε, πηγαίνει στι κατοχώρε για να εξηγήσει τον Πρωθυπουργό της χώρας ε, μερικά πράγματα για την Ελλάδα, πράγμα το οποίο βρίσκω πάρα πολύ θετικό εκ μέρους του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την έκθεση. Και θα ήθελα να ήσασταν πιο φιλόδοξος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ φιλόδοξη. Αυτό είναι και ίσω ο λόγο για τον οποίο μου αρέσουν αυτοί οι οδικοί χάρτε. Γιατί είναι πολύ φιλόδοξα έργα. Και πρέπει στα σοβαρά πιστεύω να ρωτηθούμε πώ θα επιτύχουμε του στόχου που ορίζονται ε, σε αυτού του οδικού χάρτε. Α ε, ε, φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη σα. Ο στόχος λοιπόν είναι να περιοριστεί στο ίμιση μέχρι το 2030 η χρήση των ε, αυτοκινήτων και να εξελιχθεί εξ ολοκλήρου μέχρι το 2050 στα αστικά κέντρα. Δηλαδή να μην υπάρχουν βέβαια αυτοκινήτων με παραδοσιακά καύσιμα. Να μην υπάρχουν αυτοκίνητα παραδοσιακά καύσιμα μέσα στις ε, πόλεις και ε, στο 40% μέχρι το 2050 να πέσουν τα, η χρήση των παραδοσιακών καυσίμων στην αεροπλοεία. Αυτά δεν είναι μικρά βήματα, εδώ μιλάμε για επαναστατικά μέτρα. Και καλό είναι αυτό, χρειάζομαστε μια επανάσταση στον χώρο των μεταφορών, όπως ακριβώς τι χρειαζόμαστε και στον ε, τομέα που συστούσαμε νωρίτερα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Για να είμαστε επαναστάτες λοιπόν, χρειάζεται περισσότερη καιροτομία, έρευνα, ανάπτυξη. Αυτό θα έχει κρίσιμη σημασία για την, ε, για την επιτυχία του οδικού χάρτη. Και είναι άκρο σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν το πράξουμε, ας είμαστε κεραριστές, σε 20-30 χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι να οδηγούμε τα ενδικά, τα κινέζικα, τα βραζιλιάνικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν δεν το κάνουμε εμεί δηλαδή, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι και θα αγοράσουμε εμεί τα δικά του αυτοκίνητα. Όπω τώρα, Φερρυπίν, ε, η πολιτεία τη Καλιφόρνια τη Πολιτείε ε, αναλογίζεται το ενδεχόμενο να αγοράσει ε, ηλεκτρικά τρένα υψηλή ταχύτητα, όχι από την Ευρώπη, αλλά από την Κίνα. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε μπροστά μα. Καλό λοιπόν ο δικό χάρτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλό ο δρόμο, καλή επιλογή, με την βασική ε, αρχή του ότι ο χρήστη πληρώνει, ο ρηπαίνων πληρώνει, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτέ τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να εσωτερικευτεί το εξωτερικό κόστο, πιστεύω, πράγμα το οποίο έχει κρίσιμη σημασία. Και επιπλέον αυτού, για να καταστεί δυνατό ο πραγματικό ανταγωνισμό, χρειάζεται εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστου και, κόστους και επίση θα πρέπει να δούμε Είναι. Νέες καθαρές προκλήσεις μεγάλης λοιπόν ε, σημασίας Για τους δρόμους μας. από αυτό. Όχι, είναι αστείο. Και έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από την ε, ε, από την εσφαλμένη επιλογή της επιδότησης των, ε, της υποστήριξης των ε, ορυπτών καυσίμων που θα ήταν εσφαλμένη λύση. Και Πρόεδρε παρακαλώ να, συζητήσετε και με τον κύριο Σκυλακά και τον Αρθιό όταν επιστρέψει λένε. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Οι τροπολογίες σας και οι τροπολογίες των συνοδέλφων σας είναι ευπρόσδεκτες και θα εμπλουτίνουν ασφαλώς την έκθεση. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόπουλος και ύστερα από εκείνον ο επόμενος ομιλητής, ε, επόμενη ομιλήτρια κυρία Ρόσπαχ Κύριος Τρεμόπουλος τώρα. Πρόεδρε, θα σας μεταφέρω και εγώ κάποιες πρώτες σκέψεις ως ε, σκιώδης συγητής από τη μεριά των ε, πράσινων για αυτή την αιτιολογημένη γνώμη. Καταρχάς, μια μείωση 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 συνολικά από τον κλάδο των μεταφορών δεν είναι ένας αρκετά φιλόδοξος στόχος για την προστασία του κλίματος. Αλλά τουλάχιστον αυτός ο στόχος πρέπει να καθοριστεί με τον πιο δεσμευτικό τρόπο. Οι στόχοι για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στις οδικές μεταφορές αλλά και στις αεροπορικές και την αυσιπλοεία υπολείπονται σαφώς του προσδοκομένου. Πρέπει άμεσα να βρούμε τρόπους για τη μείωση των μετακινήσεων και των μεταφορών, όχι για την αύξησή τους που προτείνει έμεσα η Επιτροπή. Καθώς και να γίνει μετάβαση σε πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους κινητικότητας. Η αρχή οριπέρων πληρώνει πρέπει να εφαρμοστεί όπως και η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γραμμή της Κομισιόν, αλλά δίνοντας έμφαση σε μερικές από τις πτυχές. Σε άλλες στεκόμαστε επιφυλακτικοί. Για παράδειγμα, στο θέμα των, του σιδηροδρόμου. Τι γίνεται στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Να σας πω από την Ελλάδα, η εμπειρία μου είναι ότι η Τρόικα, η Κομισιόν καταργούν τα δύο τρίτα των σιδηροδρομικών γραμμών. Τι σχέση έχουν όλα αυτά, αυτές οι πολιτικές, με αυτά που συζητάμε. Θα πρέπει λοιπόν η πλειοψηφία, αν όχι όλες οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατευθυνθούν προς τη σιδηροδρομική υποδομή και την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Όχι στην κατάργησή τους και μάλιστα παραβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επιπλέον, η χρέωση των φορτηγών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και η αποδοτικότητα στην κατανάλωση των καυσίμων των υπερβαρέων οχημάτων θα πρέπει να αριθμιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως συμβαίνει με τα επιβατικά οχήματα. Οι περιοριστές ταχύτητας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για τα φορτηγά για παραπέρα μείωση των εκπομπών και βελτίωση της ασφάλειας. Για τα βιοκαύσιμα. Οι ισχύοντες κανόνες δεν παίρνουν υπόψη τις μεταβολές των εκπομπών από την αλλαγή των χρήσεων γης λόγω της μετατόπισης στην παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή αυτό που λέμε τις έμεσες εκπομπές από τη χρήση γης. Μέχρι να ληφθεί πλήρως υπόψη η ισορροπία στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα βιοκαύσιμα δεν συμβάλλουν περισσότερο στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή από ότι τα ορυκτά καύσιμα τα οποία υποτίθεται ότι αντικαθιστούν τα βιοκαύσιμα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις βιώσιμες μεταφορές μόνον αν ο τομέας γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός και μειώσει τη συνολική ανάγκη για καύσιμα. Και εφόσον τα κριτήρια βιωσιμότητας αλλάξουν για να ενσωματώσουν το σύνολο των κλιματικών επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των έμεσων εκπομπών από τη χρήση γης. Για τη διεθνή ναυτιλία οι εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν άμεσα. Οι διεθνείς συνομιλίες δεν μπορούν να προχωρήσουν μέχρι ότου οι περιφερειακές οικονομικές ομάδες ρυθμίσουν τις εκπομπές του κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κρατήσει μια ανοιχτή στάση σε ό,τι αφορά ένα διεθνές σύστημα για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων από τα πλοία και να μην επιμείνει σε μέτρα που αφορούν μόνο το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια ναυτιλία. Η απόφαση έχει ήδη πάρθει για την εισαγωγή της ναυτιλίας στους στόχους μείωσης εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013, εφόσον ένα διεθνές σύστημα δεν έχει καθοριστεί ως το τέλος του 2011 και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ταχύτατα. Τέλος, η φορολόγηση της κυροζήνης έχει ήδη καθυστερήσει και ο συνολικός αντίκτυπος των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί προκειμένου να σχεδιαστούν πιο αποτελεσματικά τα συστήματα διαχείρισης πτήσεων. Με αυτές τις παρατηρήσεις ευχαριστώ και κλείνω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρεμόπουλε. Και τώρα θα λάβει τον λόγο η Χάνα Ρόσμπαχ. Η επόμενη Γκρότε Πρόντι και Σόφι Κόνη. Παρακαλώ. Τώρα η κυρία Ρόσμπαχ. Πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συζητούμε τις επιδόσεις και τα θέματα ενέργειας για το μέλλον και αυτό ιδιαίτερα συνδέεται με Εντάξει, για αυτές τις συζητήσεις, ε, αυτά τα οποία αναφέρουν οι συνάδελφοι αναφέρονται περισσότερο στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί για τη δική σας γνωμοδότηση. Θα ήθελα να επανέλθω στη δική σας γνωμοδότηση αντί να συζητάμε συνεχώς για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι στο 10 τι αναφέρετε εσείς. Αναφέρετε στο 10 ότι υπάρχει μαζική μετάθεση προς τις νέες τεχνολογίες. Και λέτε ότι αυτό απαιτεί χρόνο και είναι χρονοβόρο. Και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικέ καταστάσει που αντιμετωπίζουν τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Εγώ θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι στα κράτη-μέλη που δεν έχουν πλήρω αναπτύξει υποδομέ θα αποφασίσουν ίσως να μην συνεχίσουν τις παλαιάς τεχνολογίας μεταφορές και να περάσουν να κάνουν ένα άλμα αμέσως ε, στο μέλλον αλλάζοντας τα πάντα. Αυτό θα σου έδινε μεγάλο προτέρημα όσον αφορά α, τις συγκεκριμένες ανάγκες μεταφορών. Θα ήθελα να επανέλθω στο έγγραφό σας. Με εκπλήσει κάπως το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές κάπως αγνοήθηκαν ή αμελήθηκαν μου φαίνεται ότι είναι μια, ένα θέμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Το ίδιο αφορά και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές στην Ευρώπη και τα τρένα υψηλής ταχύτητας και για τη μεταφορά επιβατών και αγαθών. Δεν είναι κάτι στο οποίο έχετε επικεντρωθεί με ιδιαίτερο τρόπο επαρκώς. Το ίδιο ισχύει και μπορεί να εφαρμοστεί και για τα τρένα για την αντικατάσταση μικρών αποστάσεων πτήσεων μέσα στα ίδια τα σύνορα της επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχετε παρκώς λάβει υπόψη αυτά και σίγουρα θα έπρεπε να προβλέψουμε να δούμε την ανάγκη κατάθεσης μιας τροπολογίας επ' αυτών. Επίσης, για αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σε σχέση με την γνωμοδότησή σας, γενικά δεν αναφέρεται, δεν αναφέρεται καθόλου ποσοστά καθόλου μόνο στο τέλος τέλος κάνετε κάποιο λόγο για συν ή πλην 10% όσον αφορά τα καύσιμα. Ελπίζω ότι επικεντρωνόμενος στα θέματα αυτά θα καταφέρετε, θα καταφέρουμε στο τέλος να είμαστε επαρκώς θαραλέοι και γενναίοι, να καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ως πρωτοπόροι και να φτάσουμε εκεί που βρίσκονται οι Κινέζοι και να κινηθούμε προς τα εμπρός. Δηλαδή κινητήρες με μπαταρίες, με συσσωρευτές, αντί να κάνουμε μικρά μικρά βηματάκια, θα έπρεπε να έχουμε το θάρρος να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς κάτι το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο π.χ. στην Κίνα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρόσπαχ για την παρέμβασή σας και για το φιλόδοξο θα έλεγα τρόπο με τον οποίο αν διατυπώθηκε η παρέμβασή σας για φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές. Και περνάμε τώρα στις άλλες παρεμβάσεις, στους υπόλοιπους αγορητές. Ο κύριος Γκρότε, ο επόμενος αγορητής. Μετά ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θερμά συγχαρητήρια για την σύνταξη αυτή τη γνωμοδότηση, τη γνωμοδότηση αυτή. Όταν στον τομέα μεταφορών θέλουμε να πετύχουμε πραγματικά κάτι, αν θέλουμε να πορευθούμε προς την σωστή κατεύθυνση, δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε, να εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος. Και αυτό το σύστημα εσωτερικεύσης των εξωτερικών κόστων να μπορέσουμε να το διευρύνουμε και να το καταστήσουμε το μόνιμο σύστημα. Δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιες προβλέψεις ε, εφιαλτικές ότι οι ανταγωνιστές από την Άπο Ανατολή θα μας ξεπεράσουν και θα μας αφήσουν πίσω. Αν έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κοινοτικό σύστημα εσωτερήκευσης των εξωτερικών κόστων, τότε δεν διακινδυνεύουμε τίποτα. Εσωτερικοποίηση, εσωτερήκευση των, εξωτερικο, των εξωτερικών δαπανών. Μια έντιμη σωστή κάλυψη και αντιμετώπιση όλων των συστημάτων μεταφορών. Και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σωστό. Σημαντικό είναι επίσης σε αυτή την έκθεση να αναφέρουμε αυτά τα οποία αφορούν τα αστικά κέντρα αλλά και τις περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Έχουμε διαστρωμάτωση πολυμερή και ποικιλόμορφη και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Να δούμε τις διαφορετικές καταστάσεις που πρέπει να τις εξετάσουμε και να τις αξιολογήσουμε. Πώς περιφέρειες σε μία αστικά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να μετακινούνται οι πολίτες εκεί, να φτάνουν στο χώρο απασχόλησής τους και τις δημογραφικές αλλαγές να λάβουμε επίσης υπόψη. Αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό και δεν υπάρχει σε αυτή τη γνωμοδότηση ότι όλα τα σημεία σε μια τέτοια συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις κλιματικές αλλαγές να τα λάβουμε υπόψη ότι αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε και αν θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο ανταγωνισμού και προστασίας των φυσικών πόρων αλλά και αποτελεσματικότητας να έχουμε και μία μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων. Αν αυτά τα μέτρα που εγκρίνουμε και αποφασίζουμε είναι φιλοκοινωνικά, είναι κοινωνικά εφικτά και δυνατόν να λειτουργήσουν και μπορούν να συνεισφέρουν στην κινητοποίηση των πολιτών. Θα συνεισφέρω με τροπολογία και από πλευρά τη κυρία Αγιάλα Σέντερ αναφέρθηκε ο τομέα των μεταφορών να ληφθεί υπόψη. Όλο και περισσότερε μεταφορέ θα έχουμε. Αυξάνονται οι μεταφορέ στο εύρο του και είναι λογικό γιατί σε αυτόν τον πλανήτη όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν και έτσι θα πρέπει να λάβουμε όλες αυτέ τι πτυχέ στις επόμενες δεκαετίες ε, και να λάβουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό κοινωνικές επιπτώσεις σε μελέτες <clears throat> εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και να μην έχουμε φόβους ότι θα καταστραφεί ο κόσμος και θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, θα έχουμε καλές συνταγές και θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ πραγματικά. Ο κύριος Πρόντι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω γύρω από δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα των συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς, δηλαδή η φροντίδα του interface των διαφόρων ε, τρόπων μεταφοράς ε, μεταξύ σιδηροδρόμου και αστικών συγκοινωνιών, όπως επίσης ε, και την φροντίδα για τα μέσα εκείνα τα οποία εξοικονομούν ακόμη περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγμα τα ποδήλατα, μιλάω εδώ για τη δημιουργία ποδήλατοδρόμων κλπ. Θα ήθελα να κάνω επίσης μία ανοίξη προς την υποχρέωση που έχουμε να θεωρήσουμε τις μεταφορές όχι απομονωμένες μεταξύ τους αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης της κοινωνίας μας και εξηγούμε Εξηγούμε εδώ με ένα παράδειγμα. Η οικοδομική αγορά αφέθηκε ελεύθερη με δυνατότητες κερδοσκοπίας, αύξησης των τιμών, Θα πρέπει κατά συνέπεια να φροντίσουμε οι μεταφορές να μην είναι αυτές οι οποίες θα χρεώνονται την κερδοσκοπία στον οικοδομικό τομέα. Τι θέλω να πω. Πολλές περιοχές ε, ακριβένουν και αυτές αυτή η ακρίβεια μετά φορτώνεται στον τομέα των μεταφορών. Αν καταφέρουμε να χτίζουμε κατοικίες κοντά στους χώρους εργασίας, μειώνουμε και το κόστος μεταφοράς. Επίσης, Με τον Γαλιλαίο μπορούμε να έχουμε και το road pricing, να φορτώνουμε το κόστος των μεταφορών με το πραγματικό κόστος του για την κοινωνία και για το άτομο. Και αυτό για να εντάξουμε τις μεταφορές στο γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης των υποδομών μας. Ευχαριστώ, Βιτόριο Πρόντι. Ο κύριος Ρίχα Ζέμπερ έχει τον λόγο, παρακαλώ. και μετά τα ταρέλα. Ο κύριος ε, Σέιμπερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν συζητάμε για θέματα μεταφορών, θα πρέπει χωρίς ιδεολογικά προκατηλημένες απόψεις να συζητούμε. Και ως πολιτικοί πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά, να λειτουργούν σωστά οι μεταφορές. Και νομίζω ότι και οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι πολιτικές και οι πολιτικοί χωλένουν και τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Θα πρέπει να αλλάξουν αυτά και να υπό τον όρο ότι θα είναι λειτουργικά και θα λειτουργούν. Δεν θα πρέπει εδώ με απαγορεύσεις να ξεκινήσουμε. Λάθος πολιτική θα είναι αυτή. Και ας λάβουμε υπόψη μια πόλη σαν τις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί κανείς να περιορίσει τις μεταφορές και τη μετακίνηση με αυτοκίνητα και σε σχέση με την, τις υποδομές χωρίς να έχει διευρύνει τις υποδομές για τα τράμα, τον υπόγειο κτλ. Εδώ λοιπόν το δημόσιο καλείται να δράσει, να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, η εσωτερικοποίηση των εξωτερικών κόστων είναι σημαντικό θέμα. Όχι μόνο για τις ροές των μεταφορών, αλλά και για τις δυνατότητες επενδύσεων και της χρηματοδότησης των υποδομών και των αναγκών ώστε να έχουν οι πολίτες την δυνατότητα να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους ε, που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό οι πολίτες, πρέπει όμως να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις για να το κάνουν. Δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα πολύ αναποτελεσματικό σύστημα σιδηροδρόμων. Παρότι αποφασίσαμε ένα σύστημα απελευθέρωσης ε, των σιδηροδρόμων, εξακολουθούν να υπάρχουν εθνικά συστήματα σιδηροδρομικά και σε αυτά σκέφτονται τα κράτη-μέλη. Από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Βιέννη ή το Ίνσμπρουκ ε, να αγοράσει κανείς ένα εισιτήριο για να το πάρει κανείς ε, πρέπει να ακολουθήσει κλασικές μεθόδους ε, και δεν έχουν εξυγχρονιστεί τα συστήματα. Εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε με την οτροπία των κρατών μελών στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και από το Βόρειο Τυρόλο στο Νότιο Τυρόλο, από την Αυστρία στην Ιταλία δηλαδή, υπάρχουν δυσκολίες και όσον αφορά από την Αυστρία με τους Ιταλούς. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά τα προβλήματα να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν. Και έχει δίκιο ο Γκρότε όταν λέει ότι πρέπει κοινωνικά να υπάρξουν οι μελέτες των επιπτώσεων. Δεν πάνε για πλάκα, δεν κάνουν αυτές τις διαδρομές οι πολίτες για πλάκα, πάνε στη δουλειά τους. Και όταν πάνε στη δουλειά τους δεν είναι δυνατόν να μένουν επί ώρες ε, μέσα στις ε, ε, ουρές που δεν μπορούν να κινηθούν. Εδώ λοιπόν έχει πολλή δουλειά να κάνει ο πολιτικός κόσμος. Αλλά καλό χωρίς ιδεολογικούς φραγμούς ε, και περιορισμούς ε, με πραγματιστικό ρεαλιστικό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ που μας επεσήμανε τόσο σημαντικά θέματα μονοπόλια παραδείγματι στον χώρο των μεταφορών και ιδιαίτερως στους σιδηροδρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Τακταρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν εμείς θέλουμε μια ανταγωνιστική και αηφόρο πολιτική μεταφορών, θα πρέπει να μαζικά να επενδύσουμε στην υποδομές και στην ε, συνδυασμένες μεταφορές. Εγώ για να έρθω στο Στρασβούργο πρέπει να πάρω αεροπλάνο στον Πάρη, να κατέβω στη Ρώμη, από τη Ρώμη στη Μασαλία και μετά από τη Μασαλία ένα άλλο αεροπλάνο για να φτάσω στο Στρασβούργο. Για να φτάσω πιο γρήγορα γνώρισα τους ελβετικούς σιδηροδρόμους που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εμείς αντιγράφαμε τις συνδυασμένες μεταφορές ε, και τους ελβετικούς σιδηροδρόμους θα βρίσκαμε λύσεις. Εγώ παίρνω το αεροπλάνο από τον Μπάρι, φτάνω στη Ζηρίχη και από εκεί με το τρένο έρχομαι στο Στρασβούργο. Και είναι η καλύτερη λύση εντυπωσιάστηκα από τις συνδυασμένες μεταφορές της μικρής Ελβετίας. Εγώ είδα σιδηροδρόμους, ανοιχτούς σιδηροδρόμους που φτάνουν στο κέντρο της πόλης και κατεβαίνοντας από το τρένο βρίσκει κανείς το μέτρο, το ταξί, το πούλμαν, το κτέλ, τα πάντα. Λειτουργούν τα πάντα με ελβετική όπως λέγεται ακρίβεια. Ένα άλλο παράδειγμα Μιλάμε μια μέρα παραμέρα εδώ τουλάχιστον για το διοξίδιο του άνθρακος και τη μείωσή του. Λοιπόν, σκεφτήκατε εσείς ποτέ τι συμβαίνει με τα πλοία που περνάνε το κανάλι του Σουέζ, τι τραβάνε μέχρι να φτάσουν στο Ρότερνταμ. Γιατί η Ευρώπη, δεν λέω η Ιταλία, δεν κατάλαβε ότι μπορούμε να μειώσουμε κόστος, ωράρια, εργασίας, φανταζόμενοι ένα άλλο Ρότερνταμ στο κέντρο της Μεσογείου. Αυτό το Ρότερνταμ είναι το πρώτο λιμάνι, το πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι που βγαίνει, όταν ένα πλοίο βγαίνει από το, από το Σουέζ. Αλλά το πρώτο λιμάνι όμως, το πραγματικό λιμάνι που θα συναντούσε ένα πλοίο στην Ευρώπη, είναι το, βγαίνοντας από το Σουέζ, είναι το λιμάνι του Τάραντο, το οποίο θα, πρέπει, θα έπρεπε να είχε γίνει σαν το Ρότερνταμ. Τα λόγια μας πρέπει να γίνουν έργα και μόνο έτσι θα έχουμε μεταφορές πιο ανταγωνιστικές και πιο αηφόρες. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν δώσω το λόγο σε εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Σαντομάντο για την ακρίβεια, θα... Ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Επεσκέφθην το Παλέρμο σε μια, σε μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πρόσφατα, όπου διαπίστωσα ότι όταν είχε κανεί επιφασίσει στο τρένο δεν είναι δυνατόν πλέον να αγοράσει εισιτήριο. Μάλιστα, με προειδοποίησαν ότι ε, δεν επιτρέπεται να ανέβω στο τρένο χωρί εισιτήριο και ότι αν το κάνω θα πρέπει να πληρώσω και πρόστιμο. Και χρειάστηκε να γυρίσω πίσω τρέχοντα στο ε, γκισέ. Είχα τρία λεπτά περιθώρια μέσα στα οποία κατάφερα να αγοράσω εισιτήριο, αλλά υπάρχουν και πιο απλέ διαδικασίε. Και νομίζω ότι μπορούν αυτό να, το, ε, ε, να τις επιλέξουν αυτές τις διαδικασίες οι χώρες για να κάνουν πιο εύχριστες τις ε, μεταφορές. Ο εκπρόσωπος Επιτροπής παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για τα όσα είπε, για τις παρατηρήσεις του. Έχουμε μπορώ να πω, ενθαρρυνθεί στις προτάσεις μας για τη συνέχεια και την πορεία προς τη Λευκή Βίβλο. Στη Λευκή Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει στόχο για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050 κατά 60% αλλά και ε, μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο στο μισό και το, την περιστολή της αυξανόμενης ε, κυκλοφοριακής συμφόρησης. Φιλόδοξη στόχη, πολύ φιλόδοξη στόχη όχι που δεν θα πρέπει να επιδιωχθούν με τη λύση του περιορισμού της κινητικότητας, γιατί αυτό θα ήταν εις βάρος και της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι άλλες πτυχές να διερευνηθούν στο επακρό πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα περισσότερα από τα πράγματα που ε, υπάρχουν ε, καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας, γνώση των τρόπων μεταφοράς, του συνδυασμού, καλύτερη επιμελητία. Και μαζί με το φιλόδοξο στόχο 2030-2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προτείνει μια σειρά από πρωτοβουλίες, εκ των οποίων πολλές ή κάποιες είναι εξίσου φιλόδοξες με τους στόχους αυτούς όπως η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως η διαμετακόμιση, η οδική διαμετακόμιση στα λιμάνια, όπως η του ιστορικού κόστος, όπως η δημιουργία ενός δικτύου λιμένων, πολυλειτουργικού και με βάση τους ε, διαδρόμους, όπως ο περιορισμός των στρεβλώσεων στη φορολογία και ελπίζουμε έτσι πώς το Κοινοβούλιο θα στηρίξει τις φιλόδοξες αυτές τις πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι με αυτά μπορώ να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν όμως... Έχω μια ερώτηση. Στο πλαίσιο της εργασίας στην Επιτροπή ε, προβλέπετε να χρηματοδοτήσετε δίκτυα μεταφορών για τις μεταφορές με φορτηγά, να στηρίξετε αυτές τις μεταφορές. Επί παραδείγματι ε, αυτοκινητοδρόμων μέσω αυτο... αυτοκινητοδρόμων υπάρχει να προχωρήσετε σε αυτή τη λύση και σε ποιο βαθμό θα τη στηρίξετε ως Επιτροπή. Απάντηση. Η πρόταση για τη χρηματοδότηση... Η πρόταση αυτή για την χρηματοδότηση του δικτύου μεταφορών, των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών σε σχέση με την ημερομηνία της της 19ης Οκτωβρίου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής της απόφασης θα εξετάσει τη δημιουργία ενός συντονισμένου συστήματος ευρωπαϊκών μεταφορών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά εκείνου του συστήματος που θα ταυτοποιεί προτεραιότητας διαδρόμους και εγχειρήματα και σχέδια και προγράμματα. Μέσα σε αυτά θα δοθεί προτεραιότητα σε εκείνα που έχουν, πώς να το πω, είναι πιο ευνοϊκά για την αηφορία όσον αφορά τις μεταφορές είτε με άλλο τρόπο δηλαδή θα είναι η προτεραιότητα σε σιδηροδρόμους, είτε στην ε, αντιμετώπιση στενοπών ε, και προβλημάτων ή δημιουργία διευκολύνσεων, διευκολύνοντας τις πολύτροπες ε, ποικιλόμορφε μεταφορές και την χρήση επίσης των εσωτερικών ποτάμιων μεταφορών. Ευχαριστώ. Dziękuję Σας ευχαριστούμε πολύ καλά, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αισιόδοξη προσέγγιση και το αισιόδοξο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Ζέμπερ αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, μία ερώτηση θα είχα προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποθέτω ότι είναι από την Γενική Διεύθυνση Τραν Μεταφορών. Πώς λειτουργεί η συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης για το κλίμα, κλίμ, και για την Γενική Διεύθυνση Τραν Μεταφορών. Ποια είναι η συνεργασία σας και ποια είναι η προσέγγιση όσον αφορά τις αστικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε τον λόγο εκπρόσωπε της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος. Λοιπόν, πράγματι τώρα η πρώην Γενική Διεύθυνση Τραν Μεταφορών έχει χωριστεί στις, ε, στην Γενική Διεύθυνση ε, Τραν και ε, μεταφορών δηλαδή και ενέργειας και όσον αφορά την, την προετοιμασία του οδικού χάρτη με την Γενική Διεύθυνση Κλίματος και για τον οδικό χάρτη και την ε, δράση μας βασιζόμαστε σε αυτό το σενάριο. 60% μείωση των εκπομπών ρήπων για τις μεταφορές που προέρχεται από μια κοινή προσέγγιση προτύπου που έδειχνε ότι αυτό τι είναι η πιο αποτελεσματική στοχοθέτηση για την δραστηριοποίησή μας σε σχέση με τη συνολική στρατηγική μας. Αυτή είναι η απάντηση σε, αυτό το, σε αυτή την παρέμβαση, την πρώτη ερώτηση. Για τη δεύτερη παρέμβαση, τη δεύτερη ερώτηση για τις αστικές μεταφορές. Στην Λευκή Βίβλο έχει δοθεί με εμφαντικό τρόπο ε, η κάλυψη των αστικών μεταφορών, διότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ε, ε, φιλόδοξη συνολική στοχοθέτηση δεν θα ήταν δυνατόν να αγνοήσουμε τη σημασία σημαντική αναλογία τμήματος μεταφορών που καλύπτεται σε μικρές αποστάσεις, μικρές ε, κοντινές αποστάσεις μέσα στα αστικά πλαίσια. Προφανώς η Λευκή Βίβλος δεν είναι πρόγραμμα αποκλειστικά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά. Νομίζουμε ότι έτσι έχουμε δώσει την δυνατότητα να παρέμβουν και οι τοπικές αρχές, δήμοι, κοινότητες και υπάρχει ανάγκη η επικουρικότητα να λαμβάνεται υπόψη επίσης στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Ελπίζουμε ότι παρέχουμε τα μέσα και τα εργαλεία που σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να χρησιμοποιηθούν και να είναι χρήσιμα όπως ελπίζουμε ώστε να ακολουθηθεί αυτός ο τελικός στόχος, ο απότερος στόχος και η επίτευξή του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε εκπρόσωποι της Επιτροπής και αυτό ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο αυτό το σημείο που είχαμε στην ημερήσια διάταξη για αυτό το θέμα. Και τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω απλά ότι την 11η Οκτωβρίου Μέχρι τότε μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Αυτή είναι η καταληκτική προθεσμία, η 11η Οκτωβρίου. Η ψήφιση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΕΝΒΗ προβλέπεται στις 27 Οκτωβρίου και στην Επιτροπή Τραν Μεταφορών στις 22 ε, Οκτωβρίου. Ενθαρρύνω να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι τότε που θα εμπλουτίσουν σίγουρα αυτή τη γνωμοδότηση και θα την καταστήσουν πιο αποτελεσματική. Περνάμε τώρα στη συνέχεια στο επόμενο σημείο μας, στην ημερήσια διάταξη, που είναι το σημείο 16. Με άλλα λόγια, η παρουσίαση μιας μελέτης για την επιρροή όσον αφορά την εξόριξη του σχιστολιθικού αερίου και την εκμετάλλευση του, του σχιστολιθικού αερίου και τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ήμουν εγώ ένας από εκείνους που ήταν σε σχέση με τη συζήτηση αυτών των θεμάτων όταν γνώρισα, έμαθα για μια μελέτη που τον Ιούλιο είχε προετοιμαστεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Πολιτικών, σκέφτηκα ότι ήταν μια σκανδαλώδης περίπτωση πολύ μονομερής ε, ήταν ένα κομμένο και ραμμένο εγχειρίδιο για τους αντιπάλους του σχιστολιθικού αερίου. Πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι η εξόριξη στην Ευρώπη θα αναχαιτιζόταν, θα σταματούσε ώστε να μην μπορέσει να ε, θεωρηθεί ε, κάτι βιώσιμο οικονομικά και κερδοφόρο. Αυτό με κάνει να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις, κάποια ερωτήματα. Γιατί το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε τέτοιου είδους ε, μελέτες να ε, προετοιμάζονται με το δικό μας έμβλημα στο, στις εξωσελίδες και στις μέσα σελίδες να αναγνωρίζει κανείς με τα ε, ψηλοτυπωμένα γράμματα ότι δεν ήταν δική μας αυτή η παρέμβαση ή συμβολή θα πρέπει να μας βοηθήσει να αποφύγουμε τέτοιου είδους συγκρούσεις σε μελλοντικέ μελέτες και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι αντικειμενικές αυτές οι μελέτες ώστε ή να αποφεύγονται ε, τέτοιου είδους συγκρουσιακά σημεία. Δεν μπορεί η διοίκηση του Κοινοβουλίου να εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο και να δεσμεύεται με μια τέτοια μελέτη σαν αυτήν και να αναφέρεται στη συζήτηση αμέσως ποιες είναι οι μονομερείς θέσεις ε, και οι προκατηλημένες ε, τοποθετήσεις ουσιαστικά από πλευρά της διεύθυνσης των εσωτερικών πολιτικών θα πρέπει να ζητηθούν ευθύνες και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για το πώς καταλήξαμε σε αυτή τη μελέτη. Στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να παρέμβω στη συζήτηση που θα διεξαγάγουμε. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση και ο πρώτος αγορητής θα είναι... Ένα λεπτό. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο θα είναι ο κύριος Ματίας Αλτμαν και από την ομάδα επιστημόνων που ήταν αρμόδιοι για την, την σύνταξη αυτής της μελέτης και μετά έχουμε και άλλους ε, που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Έρχομαι, έρχομαι, θα φτάσω και σε αυτό. Θα αναφέρω όμως πρώτα αυτούς που έχουν εγγραφεί για τη συζήτηση. Μακέβαν, Χιούμπνερ, Μπέιλι, Στρέγια Πρόντι, Εκχάουτ, Κολάρσκα, Κατσέφσκα και Μπαλτσίνκεβιτς. Α, και ο κύριος Αρσένης. Σιμάνσκι, Σιπ. Ε, vous m'inscrivez quelque part. Alors, je, euh, Pardon, Τι λέτε κύριε Σιμάνσκι? Ευχαριστώ. Θα πρότεινα να παρουσιάσουμε τις θέσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καρουσέλ εκ περιτροπής παρεμβάσεων των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων ως ήθιστε. Η κυρία Μακάβαν λοιπόν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ζήτησα το λόγο, Είχατε, είχετε δώσει το λόγο σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι έχουμε ζητήσει από, από πλευρά στον συντονισμό τον αυτή την ε, συζήτηση. Εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε με τα συμπεράσματα της της μελέτης που είναι ανεξάρτητη μελέτη. Έχουμε όμως εδώ την παρουσίαση της έκθεσης και αυτό έχουν ζητήσει συντονιστές από τη γραμματεία. Αυτό έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ πέρα, γι' αυτό σας παρακαλώ να ακούσουμε την έκθεση πρώτα. Και βεβαίω και είχαν κάθε δικαίωμα οι συντονιστές να ζητήσουν αυτή τη μελέτη. Μα ήδη το είπαμε ότι ο κύριος Άλτμαν θα μιλήσει πρώτος. Και ο οποίος εκπροσωπεί το Think Tank ε, που προετοίμασε, την ομάδα που προετοίμασε αυτό το έγγραφο. Ε, ωραία. Ας αρχίσουμε με τον κύριο Αλτμαν. και μετά συντονιστές και παρόντες σας πάρουν το λόγο. Και μετά όποιος άλλος ε, έχει εγγραφεί στη συζήτηση θα μιλήσει. Ο κύριος Άλτμαν καταρχήν. Mr. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εκλήθημε να εξετάσουμε τις συνέπειες από την εξαγωγή σχισολιστικού φυσικού αερίου τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και πιθανούς ε, ρόλους ε, που θα μπορούσε να δραματίσει το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην, ε, στο μέλλον σε μια κοινωνία, οικονομία καλύτερα απελαγμένη από άνθρακα. Μιλάμε λοιπόν για μη συμβατικό αέριο αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο το αέριο είναι μη συμβατικό. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξαγωγή του από τα βάθη της γης είναι μη συμβατικό, τρία διαφορετικά είδη δηλαδή μη συμβατικών αερίων με κύριο κοινό χαρακτηριστικό ότι συνεπάγεται σημαντική προσπάθεια ε, η εξόριξή τους από τα γεωλογικά στρώματα. Ξεκινώ λοιπόν με τις ε, περιβαλλοντικές συνέπειες και τους κινδύνους και θα λέγω ότι ο όρος κίνδυνος είναι πολύ πιο σκόπιμο να χρησιμοποιείται από τον ε, ε, όρο συνέπεια. Γιατί αυτό που μπορούμε να δείξουμε είναι ο κίνδυνος από την εξόριξη του ε, φυσικού αερίου και βέβαια να εκφράσουμε και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να έχουμε νομοθεσία που θα μας προστατέψει από τους κινδύνους. Πολλές είναι οι συνέπειες λοιπόν. Πρώτη και μία αναπαφευκτή συνέπεια, γιατί χρειάζεται πολύς χώρος, η επιφάνεια που αξιοποιείται, καταναλύσκεται κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Χρειάζεται πρόσβαση, χρειάζεται ε, σκάψιμο, χρειάζεται μεταφορά, είτε πρόκειται για αγωγό, είτε πρόκειται για μεταφορά με φορτηγά. Συνέπειες καλύτερα κίνδυνοι είναι οι εκπομπές ε, ρηπογόνων, ρήπανση των, ε, του υδάτιου ορίζοντα, υπόγειων υδάτων ή επιφανειακών, πιθανόν δε και τεράστια κατανάλωση, υψηλή κατανάλωση ε, υδάτων, πράγμα το οποίο σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως έχει αποδείξει η σχετική εμπειρία από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Και για να σας δώσω ε, επιπλέον πληροφορίες, στις ΗΠΑ Αμερικής κατά τα τελευταία 3 με 5 χρόνια είχαμε 50.000 περίπου πηγάδια ε, που άνοιξαν για την εξαγωγή ασφιστολιθικού φυσικού αερίου. Ας ότι υπάρχει επαρκή εμπειρία από την υπόθεση αυτή, ανεξάρτητες μελέτες και εκθέσεις από την, τις ε, υπηρεσίες της κρατικές που ε, μπορούν να στηρίξουν τις δικές μας διαπιστώσεις. Στην Ήδρο υδρογρογμάτωση έχουμε πολύ σημαντική χρήση υδάτων και πιθανή ε, ραδιενεργού υλικού. Στις Ηνωμένε Πολιτείε σημειώνεται παραβίαση των νομικών προδιαγραφών σε επίπεδο 2% κάθε γεώτρησης. Δηλαδή 5.000 ε, γεωτρήσεις έχουμε περίπου 500 ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Στη Γερμανία η εμπειρία που έχουμε από την υδρορογμάτωση Υπάρχει ήδη, υπάρχει μια κάποια εμπειρία. Και ε, ρήπανση των εδαφών που θα πρέπει να αποκατασταθούν. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Έχουμε επίσης ε, πιθανή ρήπανση από μεθάνιο των εδαφών, που είναι το φυσικό στατικό δηλαδή του ασβεστολιθικού φυσικού αερίου, απελευθέρωση μεθανίου και κίνδυνος εκ του εκρήξεως. Έχουμε υψηλή περιεκτικότητα σε άλλας ε, των υδάτων και πιθανή επιμόλυνση γειτονικών ε, πηγαδιών επηρεάζονται τα βαθαία στρώματα, γεωλογικά στρώματα με κίνδυνο μικροσυσμών της κλίμακας ενός έως τριών βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε να αντλήσουμε, να ε, εξαγάγουμε ασβεστοπληθικό φυσικό αέριο. Στη δεύτερη πτυχή στις ε, επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την υγεία. Η πτυχή και το ισοζύγιο σε σχέση με, την, <clears throat> με το φαινόμενο των αερίων θερμοκηπίου. Αυτά λοιπόν τα μη συμβατικά αέρια ή το μη συμβατικό αέριο είναι ασφαλώς καλύτερο για το περιβάλλον στη χρήση του από ότι ο άνθρακας. ή για να το πω διαφορετικά είναι τόσο καλό για το περιβάλλον όσο το παραδοσιακό φυσικό αέριο, το συμβατικό φυσικό αέριο. Οι πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι μια τέτοια ανάλυση, όπως αυτή που σας έκανα τώρα, ε, μπορεί να είναι ακριβής μόνο ανάλογα με την ποσότητα μη συμβατικού φυσικού αερίου που μπορεί κανείς να αντλήσει από ένα τέτοιο πηγάδι. Γιατί, Γιατί οι εκπομπές σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από την ίδια τη γεώτρηση, από τη διαδικασία της γεώτρησης. Άρα ανεξαρτήτως του πόση παραγωγή φυσικού αερίου θα έχουμε από τη το συγκεκριμένο πηγάδι γεώτρησης, ο κίνδυνος είναι ίδιος. Άρα, εάν κατά μέσον όρο έχουμε παραγωγή φυσικού αερίου, εξαγωγή, γεώτρηση φυσικού αερίου, εξίσου σημαντική με αυτή των ΗΠΑ, έχουμε ε, ταυτόχρονα και την μεταφορά, το ζήτημα της μεταφοράς ε, από την βορειοανατολική Φερρυπίν βυρία στον, στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις σχετικές συνέπειες, δηλαδή το πρόβλημα των μεταφορών και τις συνέπειες των περιβάλλον. αλλά εάν έχουμε την εξαγωγή ε, από τον ε, επιτόπου, δηλαδή από τα μεγάλα αποθέματα θέματα φυσικού αερίου, τότε βρισκόμαστε στα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα και των απομόνων διοξιδίου του άνθρακα που έχουμε παραδοσιακά και στι ΗΠΑ μέσα με τον κίνδυνο τη ανάφλεξη. Άρα, το ισοζύγιο σε σχέση με, το, με τα αέρια του θερμοκηπίου, εάν είναι χαμηλότερη παραγωγή από ό,τι έχουμε στι ΗΠΑ, μπορεί και να ανατραπεί. Άρα, αυτό που σα λέω είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται από τα γεωλογικά δεδομένα στην Ευρώπη. Πρέπει πρώτα να γίνει η ανάλυση των ε, γεωλογικών διαστρωματώσεων για να δούμε αν υπάρχει επαρκή κοιτάσματα και στη, ή μάλλον επαρκή πόροι και στη συνέχεια να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Και το άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω ήταν το εάν η Ευρώπη είναι επαρκώς ε, ε, προστατευμένη έναντι αυτών των κινδύνων από την εξαγωγή, από την εξόριξη φυσικού, ασβεστολιθικού φυσικού αερίου ή αν θα πρέπει να ενισχυθεί η νομοθεσία. Πρέπει καταρχάς να επισημάνουμε ότι και να υποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν υπάρχει οδηγία πλαίσιο για τις ε, εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας οι εξορυκτικές δραστηριότητες και θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει στη μελέτη μας και ένα χειρίδιο ε, πηγή που δίνει μια ε, κατάσταση των 43 χωρών ε, του κόσμου με, τις τους, με την ομοθεσία για την εξωτερική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι υπάρχει και τι είδου ε, νομοθετικό πλαίσιο μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται λεπτομερής ανάλυση. Αυτή η αρχική εξέταση παρουσιάζει εννέα κενά ως προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα για τη δική μας την ανάλυση και κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται με τη δήλωση επικίνδυνων ουσιών και το κατά πόσον χρειάζεται έγκριση για το κατά πόσον θα παραμένουν τα χημικά αυτά στον υπόγειο ορίζοντα, ή αν υπάρχουν μελέτες, αν υπάρχει δυναμικό και ποιο είναι αυτό το δυναμικό των ε, μονάδων ε, κατεργασίας υδάτων τόσο προς τις ποσότητες, γιατί βεβαίως ε, αν έχουμε 50.000 κυβικά ε, μέτρα νερό για κάθε πηγάδι, τότε θα πρέπει βεβαίως να γίνει κατεργασία των υδάτων που θα προκύψουν. Από... Τέλειωσε ο χρόνος μου. Α, μου έχει μείνει ένα λεπτό πολύ καλά. Και έτσι θα Έχω ένα λεπτό, περνάω στο τελευταίο θέμα. Ερώτηση. Τι υπόσχεται ενεργειακά όσον αφορά την οικονομία σε σχέση με τα μη συμβατικά μέτρα οι πόροι έχουν κατεκτήμηση υπολογιστή, δεν έχουμε καλή γνώση των πόρων, δεν έχουμε σωστή και πλήρη εκτίμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων στην Ευρώπη. Η καλύτερη δημοσίευση είναι από την διοίκηση των ΙΠΑ στον ενεργειακό τομέα και είναι μια κατεκτίμηση όσον αφορά τους ε, υδρογονάνθρακες ε, και τη γεωλογική τους εκτίμηση. Έχουμε θετική εμπειρία από τις ΙΠΑ και μπορούμε να δούμε πόσο γοργά μπορούν όλα αυτά να προχωρήσουν. Όμως μπορούμε να δούμε και ποιες είναι και οι δυσχέρειες για την Ευρώπη, συγγνώμη, που είναι πολύ διαφορετική από τη ΣΥΠΑ σε πάρα πολλές πτυχές. Θα ήθελα να τονίσω στο τέλος τέλος κάτι και αυτό είναι ότι έχουμε τους πόρους που δεν είναι ισομερός ε, διανεμημένοι ανά την Ευρώπη. Έχουμε τους υποτιθέμενους μέγιστους ε, πόρους στα αποθέματα στη Γαλλία και στην Πολωνία και όσον αφορά το πάχος διαστρωμάτωσης ε, των αποθεμάτων που αναμένεται σε σχέση με την εκμετάλλευση, την άντληση αυτού του αερίου, είναι πιο τα πιο σημαντικά ε, αποθέματα και πάλι στην Πολωνία. Και αν ε, εξετάσετε όλα τα δημοσίευματα τα οποία καλύπτουν αυτή την πτυχή όσον αφορά το μη σημαντικό αυτό αέριο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας που δημοσιεύθηκε τον Μάιο εφέτος μια ειδική έκθεση, η Χρυσή Εποχή του αερίου για ένα σενάριο των επόμενων 25 ε, επόμενων ετών όσον αφορά την παραγωγή αερίου και του μη συμβατικού αερίου στην Ευρώπη, λένε αυτές οι εκτιμήσεις ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου θα μειωνόταν κατά 1,4% ετήσια μέχρι το έτος 2035. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την Νορβηγία. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Σε ευχαριστούμε πολύ Πράγματι, ο κύριος Άρτμαν που ομίλησε εξ ονόματος των συντακτών αυτής της μελέτης ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή του. Θα δώσω την προεδρία στον κύριο Λάινεν σε ένα λεπτό. Συμφωνήσαμε ότι πρώτα θα ακούσουμε εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων και έτσι παρακαλώ με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναλάβετε πάλι την προεδρία κύριε Λάινεν. Παρακαλώ. Έχουμε πάνω από 10 που έχουν εγγραφεί, ένα λεπτό καθένας από τους αγορητές. Επαρκεί πληρέστατα, θα έλεγα. Ο Ρίχαρτ Ζέιμπερ θα ήταν ο πρώτος λοιπόν. 1,5 λεπτό. Έχουμε 15 που θέλουν να μιλήσουν. Λοιπόν, 1,5 λεπτό. Κύριε Ζέμπερ, θα είμαι σχετικά σύντομος. Από πλευρά του ΕΛΚ έχουμε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την αμεροληψία, την ανεξαρτησία των συντακτών αυτής της μελέτης. Αυτό πρέπει ακόμα να ληφθεί υπόψη και να τεθεί υπό εξέταση, διότι βρίσκονται κοντά σε κάποιους οργανισμούς και οργανώσεις και θα θέλαμε σε σχέση με αυτά τα θέματα να ακούσουμε τους ίδιους τους συντάκτες αυτής της μελέτης τι λένε σε σχέση με την έγερση αυτή της κατηγορίας. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα θα ήταν σχετικά δύσκολο να συναγάγει κανείς κάποια, κάποια αντικειμενικά συμπεράσματα. Επανειλημμένα στη μελέτη αναφέρεται ότι είναι δύσκολο να έχουμε ακριβή στοιχεία διότι και τα λοιπά η τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως στη ΣΥΠΑ και ότι αυτά τα αποθέματα είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και τα λοιπά. Για να αποκτήσει κανείς μια συνολική σφαιρική εικόνα είναι δύσκολο αυτή τη χρονική στιγμή σε αυτή τη συγκυρία. Θα ήταν πιο σκόπιμο και θα, ήταν πιο, ε, θα είχε μεγαλύτερο νόημα να συνταχθεί μια άλλη μελέτη από άλλους συντάκτες της επόμενης αυτής μελέτης και αυτό θα ήθελα να γίνει σε σχέση με την προώθηση αυτής της διαδικασίας για το σχιστολιθικό αέριο. Ευχαριστώ. Μία μελέτη μετά τη μελέτη, μετά τη μελέτη, πολλές μελέτες δηλαδή. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ή αρκετές πολλέ Η αρκετέ στην αγορα Μακάρτη παρακαλώ. Well, I mean, at the beginning of this... Στην αρχή αυτής της συζήτηση, Πρόεδρε, είχαμε το ερώτημα αν θα έπρεπε να γίνει αυτή η μελέτη ή όχι, λέει η κυρία Μακάβαν και ο Αντιπρόεδρος ε, ανέφερε ότι δεν ήταν καλό να γίνει αυτή η συζήτηση, όμως ε, είναι πολύ καλό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. Είναι μια νέα προσέγγιση και έχει ιδιαίτερη πρόκληση που θέτει και πρέπει να φτάσουμε στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βάθος. Να δούμε υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο ή όχι και αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε και όταν θα εκμεταλλευτεί μια τέτοια δυνατότητα να προστατευτούν οι πολίτες, να προστατευτούν τα αποθέματα νερού, το ε, υπεδάφιο νερό και νομίζω το να λέει κανείς να μην συζητηθεί κάτι είναι γελίο, παράλογο σε μια δημοκρατία. Ξέρω ότι υπάρχει τεράστιο λόμπι και αυτό συμβαίνει και όπου και να κοιτάξει κανείς. Υπάρχουν τέτοιοι λομπίστες. Δική μας ευθύνη είναι να νομοθετήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό συμφωνώ επ' αυτού μαζί σα. Είναι η αρχή αυτή τη συζήτηση. Θα ακούσουμε, υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ αποφα... Ε, απόψει και θα τι ακούσουμε για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Πρέπει να ακούσουμε όλε αυτέ τι απόψει. Ε. Και έχουμε αυτή την κατάσταση και στη χώρα μου θα έπρεπε να γνωρίζουν οι, άνθρω... οι πολίτε ότι εδώ υπάρχει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα ενό υπουργού, όχι τη δική μου κυβέρνηση, της, φιλελεύθερη της φιλελεύθερης συντηρητικής κυβέρνησης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και λένε ότι έχουν σταματήσει οι έρευνες ε, λόγω του ότι υπήρξε ένας ε, ε, μικρότερης εμβέλειας σεισμός που σημειώθηκε. Και όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε και είμαι ευγνώμων για το ότι ενεγράφει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το δούμε σε βάθος. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Πράγματι το Αμερικανικό Κογκρέσο έκανε μια μεγάλη μελέτη και εδώ έχουμε και το ψήφισμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη μελέτη και περιβαλλοντικέ επιπτώσεις. Οι πολίτε αναμένουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έλεγα, να καλύψουμε αυτή την πτυχή, αυτό το ζήτημα, χωρίς αμφιβολία. Και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά τη σύνταξη της μελέτης, αν θα συντάξουμε μια έκθεση εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο. Ε, Εσεί παρακαλώ στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αλλά δεν ζήτησα εγώ να παρέμβω, δεν ζήτησα να μου δώσετε τον λόγο, λέει ο κύριο Τζερμπράντι. Είσαστε όμω στον κατάλογο μου εδώ των αγοριτών. Υπέροχο. Τα πιο περίεργα πράγματα γίνονται αυτό το απόγευμα εδώ. Α, θα αφήσω το, τον λόγο να παρέμβουν άλλοι. Δεν θα παρέμβω εγώ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι ένα πολύ καλό θετικό πράγμα το ότι έχουμε αυτή τη μελέτη που συντάχθηκε. Θα ήθελα να ακούσουμε περισσότερα σε σχέση με αυτή τη μελέτη από τον κύριο Αλτμαν, Αν ακούγαμε περισσότερα, θα φοβούμαι ότι θα χρειαστεί να τα διαβάσω όλα απόψε μόνο μου. Προσβλέπω στο να ακούσουμε περισσότερα. Ο κύριο Σιμάνσκι σίγουρα ενδιαφέρεται σε αυτό, για αυτό το θέμα και θα ήθελε να παρέμβει. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ αποφάσισα να εμπλακώ περισσότερο σε σχέση με αυτή την έκθεση, διότι συμμερίζομαι και εγώ την άποψη που εκφράστηκε από πλευρά Evans, για παράδειγμα ίσως εννοεί Μακάβαν ο μιλητής και καλό θα ήταν να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να συζητηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο και θα πρέπει να μιλήσουμε για γεγονότα, για στοιχεία που είναι δεδομένα επιτόπου. Πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι μια διεργασία που πρέπει να ληφθεί έτσι υπόψη με συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι μόνο το να εξετάσουμε ποια ερωτήματα αξίζουν τον κόπο, όλα τα ερωτήματα αξίζουν τον κόπο. Τώρα πρέπει να αναζητήσουμε να εξεύρουμε απαντήσεις. Διάβασα αυτή τη μελέτη κάποιες εβδομάδες πριν και είχα πολύ σημαντικές αμφιβολίες. Παράδειγμα, οι εκπομπές μεθανίου, οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται στα πρότυπα τα οποία ισχύουν στην ρωσική υποδομή που είναι τελείως διαφορετικά από όσα υπάρχουν στην Ευρώπη. Να δούμε τι θα γινόταν στην Ευρώπη. Η διαρροή όσον αφορά τις υποδομές για μεθάνιο είναι τρεις φορές μικρότερη από ό,τι στα όσα αναφέρετε εσείς. Γι' αυτό φαίνεται ότι είσαστε προκατηλημένοι εσείς μονόπλευρα. Δεύτερον, ο τομέας ε, που πρέπει να καλύπτεται από τι υποδομέ αληθεύει ότι κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 80 οι περιοχές γεωτρήσεων ήταν μέχρι 20.000 τετραγωνικά μέτρα διότι η οριζόντια γεώτρηση δεν ήταν διαθέσιμη ως τεχνολογία. Σήμερα είναι 500 έως 800 τετραγωνικά μέτρα όλα και όλα δεν κατανοώ γιατί όταν συντάχθηκε αυτή η έκθεση αυτές οι νέες δυνατότητες πιο καινοτόμε δεν ελήφθησαν υπόψη. Φυσικά μπορεί να εξετάσει κανείς αν ο νέος αυτός τύπος αερίου θα είναι βιώσιμος και κερδοφόρος στην αγορά. Αλλά αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν όσοι εμπλέκονται στην αγορά αυτή. Δεν είναι δική μας δουλειά να προβλέψουμε και να προδικάσουμε εμείς κάτι τέτοιο. Με ξέπληξε όμως ότι η αξία της αγοράς υπολογίστηκε με στοιχεία λέει τα οποία χρησιμοποιούνται από την έννοια έναν από τους μεγάλους εμπλεκόμενους στην αγορά, μεγάλους μίζωνες εταίρους όσον αφορά την αγορά και την εκμετάλλευση στην Ευρώπη. Θα έλεγα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν επιλέγουμε ε, πηγές για την πληροφόρησή μας και την τεκμηρίωσή μας. Πιστεύω ότι αυτή η μελέτη θα έπρεπε να είχε συνταχθεί από λιγότερο προκατηλημένη ομάδα ερευνητών. Μια και ε, συντάχθηκε ε, σε σχέση με άτομα που εμπλέκονται όσον αφορά στην πηγή αυτή ενέργειας υπάρχουν μειονεκτήματα. Είναι μια μείζον πηγή εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να είναι φυσικό και ομαλό ότι δεν θα ε, αφήναμε να ετοιμάσει κάποιος ε, που εξειδικεύεται στα ποδήλατα μια μελέτη για τα αυτοκίνητα ή να ετοιμάζουν κάποιοι μια μελέτη όσον αφορά εμπορική δραστηριότητα που έχουν και να συντάσσουν μελέτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα αυτοί είναι οι ισχυρισμοί που εγώ θα ήθελα να απορρίψω όσον αφορά τα μέλη της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μπορεί να συντάξει κανείς μία μελέτη για το συστολιθικό αέριο όταν είναι ερευνητής και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχω εδώ σε σχέση με μια δημοσίευση του Αυγούστου όσον αφορά το μεθάνιο και τα λοιπά. Το μεθάνιο λέει σε 85% δειγματοληπτικά ανοιχνεύτηκε και είχαμε εδώ και σε σχέση με το εύρος αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στη ΣΥΠΑ αυτό. Η κυρία Σαντρίν Πηγέ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που προχώρησαν σε αυτήν τη μελέτη μετά από αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγγέλει τις επιπτώσεις ε, του σχιστολιθικού αερίου. Ξέρετε ότι έχουμε καμιά εξενταριάμπιες που χορηγήθηκαν ε, στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία μέσα σε μια γενική θολούρα και οι τοπικοί ε, κλεγμένοι δεν είχαν ιδέα για το υπό ποιες συνθήκες δόθηκαν αυτές οι άδειες. Η εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ανάλογα με την κατάσταση και χρειάζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ρύθμιση. Η εμπειρία που έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες μας δείχνει ότι έχουν ε, μεσολαβήσει πολλά δυστυχήματα. Εγώ πήγα στην πενσιλβάνια στις Ηνωμένε Πολιτείε για να συναντήσω διάφορους. Οι πετρολικές εταιρείε λένε ότι δεν ε, υπάρχει κανένας ε, κίνδυνος, αλλά ο πραγματικός απολογισμός είναι άλλος και στο Τέξας και στην Πενσιλβάνια γίνεται σήμερα αυτός απολογισμός και η καταστροφή είναι μεγάλη. Και οι δημοκράτες υπέβαλαν στο Κογκρέσο μία ε, πρόταση για να απαγορεύσουν την τεχνική θρηματισμού που και πρέπει να λάβουμε θέση έναντι των κερδοσκόπων και αυτών που θέλουν να προστατεύσουν ε, την ε, επικράτειά τους και να προστατεύσουν τους κατοίκους. Πλεονεκτήματα υπάρχουν, πρέπει να τα ψάξουμε βέβαια στη μελέτη για την ε, αυτο, ε, ενεργειακή ε, ανεξαρτησία, οικονομίες κλπ. Είναι σχεδόν ανύπαρκτα αυτά, δεν έχουμε πλεονεκτήματα. Και σε αυτήν τη φάση αν για ορισμένους ε, που θέλουν να αμφισβητήσουν αυτή τη μελέτη και θέλουν νέα μελέτη, μπορούν να το κάνουν, όλες οι αμφιβολίες ε, έχουν υπόσταση, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει η αρχή της πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί ε, που είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου λένε ότι ακόμη υπάρχουν σημεία που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα μορατόριου για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου και θέλω να ξέρω από την Κομισιόν ποια είναι η γνώμη της για αυτό το μορατόριου και νομοθετικές προτάσεις για την υδραυλική εξόριξη σε ευρωπαϊκό πεδίο. Και ζητώ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβει απόφαση σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Γιολάντα Χιούμπεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Προσέξτε, αυτό το έγγραφο που παρουσιάστηκε δεν φαίνεται να είναι μία μελέτη ή κάποια συλλογή τεκμηρίων με πραγματογνωμοσύνη. Πρώτον, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται εδώ είναι πράγματα τα οποία δεν θα έβρισκε κανείς σε μελέτες επαϊόντων που έχουν επαληθευθεί. Αναφέρεται ότι η ικανότητα εγκαταστάσεων τέτοιων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, θα είναι ανεπαρκής. Ξέρετε ποιο είναι το δυναμικό ανεπαρκής κοινωνική συμμετοχή. Αυτό είναι αντίθετο στοιχείο στην οδηγία. Υπάρχει κοινωνική συνιστόσα σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα. Δεύτερον, εμφαίνονται αυτά σε μία μελέτη επαϊόντων. Δεν μπορούν να, αναφέρεται, να αναφέρονται ότι εμφαίνονται, αναφέρονται. Πρέπει να έχουν επαληθευτεί από την έρευνα Μπορεί κανείς να πιστεύει ότι κάτι είναι ή δεν είναι αληθινό, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι αληθινό και ότι είναι τεκμηριωμένο. Τι είδου γλώσσα και διατύπωση είναι αυτή. Να αναμένει κανείς ότι θα μπορούσαν, λέει, might be results. Θα μπορούσαν να είναι αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι αυτή η ορολογία και οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά κείμενα. Σίγουρα όχι. Ατυχήματα. Ατυχήματα έχουμε ατυχήματα με την εξόριξη πετρελαίου. Στον κόλπο του Μεξικού για παράδειγμα. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό για το όριο 3%, 3% λέει ατυχημάτων σε ατυχήματα. Ισχυρίζεστε εσείς ότι πρέπει να υπάρχει ειδικό εντοπισμός και ταυτοποίηση προβλημάτων. Αληθεύει αυτό για κάθε και οποιοδήποτε ατύχημα. Πάντα πρέπει να υπάρχει διάγνωση του κόστους του προβλήματος, οποιοδήποτε προβλήματος. Και πιστεύω ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι όλα αυτά δεν είναι χωρίς μεροληψία, μεροληπτική αντιμετώπιση από πλευρά σας. Άσχετα αν είναι συμβατικό ή όχι, η πετρελαιαγωγή και αεριαγωγή μπορεί να είναι μια πηγή περιβαλλοντικής επιβάρησης και ατυχημάτων η όχληση που παράγεται από τον μηχανισμό εξόριξης, ηχητική όχληση. Για κοιτάξτε τι γίνεται στις κανονικές ομαλές όπως αποκαλούνται εξορίξεις πετρελαίου. Υπάρχουν τέτοιοι θόρυβοι. Μη μου πείτε λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή ηχητικής όχλησης όταν θα εξορίσετε κάτι άλλο ως προϊόν και ότι επειδή θα είναι το συστολιθικό αέριο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, σας απευθύνω έκκληση. Αν θέλετε να ληφθούν σοβαρά αυτά τα στοιχεία, με σοβαρό τρόπο, ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις και διαβουλεύσεις, τότε πρέπει να βασίζονται όλα αυτά σε μια αμερόληπτη, ουδέτερη, αντικειμενική, τεκμηριωμένη επιστημονικά έρευνα. Όπως στην Αμερική. Λέτε ότι στην Αμερική το 2012 θα υπάρχουν, λέει, μόνο αποτελέσματα. Με βάση ποια στοιχεία διατυπώσατε εσείς αυτή τη θέση και παρουσιάσατε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό το έγγραφό σας για το σχιστολιθικό αέριο, για το ότι είναι, λέει, απειλή, διότι δεν θα πρέπει, λέει, να εξορίσετε. Λέτε αφενός από τη μία πλευρά ότι τα αποθέματα, λέει, στην Ευρώπη δεν θα έχουν καμία επιρροή στο μέλλον. Κάτι δεν πάει καλά με όλα αυτά και με αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πρέπει κανείς να διαφοροποιεί μεταξύ μιας μελέτης που ταυτοποιεί και δείχνει ποια είναι τα προβλήματα και των πολιτικών συμπερασμάτων που μια χώρα, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η μελέτη δεν λέει ότι το σχιστολιθικό αέριο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δυνατότητα και να το εκμεταλλευτούμε, αλλά να δούμε ποια προβλήματα ίσως μπορεί να υπάρχουν. Αυτή ήταν η εντολή και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Η Εντίτε Στρέλα, είπα 1,5 λεπτό, είναι πάρα πολύ. Πόσοι θα λάβουν τον λόγο, από όλους αυτούς αν μακρηγορείτε εσείς. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω εδώ μπροστά μου, στα χέρια μου, αυτή τη μελέτη που ζητήθηκε από τους συντονιστές να συνταχθεί και που ζητήθηκε και από θεματολογικά να συνταχθεί όπως συμβαίνει με κάθε μελέτη. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τους ε, συντάκτες αυτού του κειμένου που βρίσκεται εκεί πάνω σε αυτό το τραπέζι που δεν έχει καμιά υπογραφή, ούτε κανένα λογότυπο ή έμβλημα. Και για να αξιολογήσω την αξιοπιστία των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται εδώ, θα ήθελα οι συντάκτες να μας αναφέρουν τα ονόματά τους, να είναι εδώ τυπωμένα τα ονόματά τους. Τούτο αυτό είναι ένα θέμα επίμαχο. Είναι ένα θέμα που αξίζει όμως τον κόπο να εμβαθύνουμε σε αυτό. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας για μία τη δήλωση ε, του 2011 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και που αφορά αυτό το θέμα, την εκμετάλλευση των σχιστολιθικών αποθεμάτων αερίου και πετρελαίου σχιστολιθικού και που παρουσιάζεται τον κύριο Ζουβά Μποβά από μένα την ίδια και από την κυρία Άννα Ρόσμπαχ. Δυστυχώς ε, ε, έληξε η προθεσμία την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θα υπάρξει καμιά πρακτική επίπτωση από αυτό. Όμως είναι σημαντικό με βάση αυτή τη μελέτη, με βάση αυτά τα οποία κάνουμε εδώ και με τις ανάγκες ε, που έχουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για το περιβάλλον και το θέμα αυτό με την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη ή με ψήφισμα ή με άλλο τρόπο να δώσουμε συνέχεια. Είναι όμως σημαντικό εμείς να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία και οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι, τι δεν πάει καλά και πάει στραβά με την εκμετάλλευση αυτής της δυνατότητας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Οι συντονιστές αύριο το πρωί το έχουν εγγράψει στην ημερησία διάταξη για την συνάντησή του Ο Βιτόριο Πρόντι τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι η μελέτη που μας παρουσιάστηκε είναι πολύ ε, λογική, επιφυλάσσομαι όμως να τη μελετήσω. Πάντως στον θρηματισμό του βράχου υπάρχει μεγάλη γεωλογική αναταραχή, διαπιστώνουμε ότι γίνονται σεισμοί, υπάρχουν απώλειες μεθάνιου και θα ήθελα να θυμίσω ότι η διάρκεια αυτών των πηγαδιών είναι πολύ μικρότερη από ότι τα συμβατικά πηγάδια. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Αν εμείς εκμεταλλευτούμε και έχω υπόψη μου την Ιταλική περίπτωση, αν εκμεταλλευτούμε τα δασικά και γεωργικά κατάλοιπα με την πυρόληση μπορούμε να παράγουμε το 1 τρίτο των αναγκών μας σε φυσικό αέριο. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε πρώτα να εκμεταλλευτούμε με το πλεονέκτημα της προσαρμογής στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών κάνοντας πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε και τα υπόλοιπα ας περιμένουμε, τα δούμε μετά. Εγώ επιφυλάσσομαι πάντως να διαβάσω τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόνεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Μαγκάβεν είπε ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει συζήτηση. Δεν ισχύει αυτό. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω καταρχά ότι η συζήτηση για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο έλαβε χώρα στι 8 Μαρτίου εφέτος στην Ολομέλεια. Και βέβαια ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Γιατί όπω είπε ο Επίτροπο Έτιγκερ στις 8 Μαρτίου, η γεώτρηση είναι αδύνατο να γίνει αν δεν την εγκρίνουν και οι πολίτες. Ωστόσο θα πρέπει και οι πολίτες να έχουν ε, αξιόπιστες πληροφορίες στη θέση τους. Και υπογραμμίζω ότι είναι μεροληπτική αυτή η μελέτη. Και είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο παρτού, ένα έτοιμο εγχειρίδιο που θα εξυπηρετήσει μόνο αυτούς που θέλουν να αποτρέψουν την εξόριξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Θα υπενθυμίσω δε ότι ο Επίτροπος Oettinger μας είχε πει ότι αποτελεί πηγή ελπίδας το συστολιθικό φυσικό αέριο. Ναι, μεν πρόκειται για ορυκτό καύσιμο, αλλά σε σύγκριση ε, ε, ως προς τον ως προς τον ισολογισμό διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ καλύτερο από τον άνθρακα ή το πετρέλαιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουράσικα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο που βλέπουμε για το συστολιστικό φυσικό αέριο. Δεν πρέπει λοιπόν να αισθάνεται κανείς ε, έκπληξη για, την, ε, για τις έντονες αυτές που ακούγονται. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση, με το που ακούγεται η πρόταση έρχεται και η αντιπρόταση για το μορατόριο. Μην ε, ξαφνιάζει λοιπόν που είναι τόσο ε, αμφισβητούμενες αυτές οι προτάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εάν η Γαλλία μετά το ατύχημα της Φουκοσίμα ε, κήρυξε μορατόριουμ στην πυρηνική ενέργεια. Και γιατί, όχι βέβαια, γιατί λοιπόν κηρύσει ε, μορατόριουμ ως προς το συστολιθικό φυσικό αέριο. Να σας πω γιατί, γιατί 80% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλία προέρχεται από την πυρηνική. Άρα η κατάσταση είναι περίπλοκη. Είναι περίπλοκη και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά και ασφαλώς αυτό σχετίζεται και με την ενεργειακή μας ασφάλεια. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όταν ετοιμάζω στο μέλλον εκθέσεις θα πρέπει αυτές να λαμβάνουν υπόψη και την πτυχή της ενέργειας και της ασφάλειας ενέργειας. Διαρκώς ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην ενέργεια και το περιβάλλον. Ενέργεια και κλίμα. Πολύ καλά. Ε, τότε λοιπόν ας γίνει μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις πτυχές της οικονομίας του περιβάλλοντος αλλά και άλλες πτυχές. Κάτι ακόμη λοιπόν και καθώς δεν είμαι ε, μηχανικός δεν πρόκειται εγώ να δώσω επιχειρήματα υπέρ κατά της υδρορογμάτωσης και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και τι θέλω να χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη κτλ. Αλλά είπατε εσείς ότι είναι για την ε, ασφάλεια, για την υγεία του ανθρώπου μάλλον ε, κακό το χιστολιθικό φυσικό αέριο και ότι είναι επικίνδυνο. Ε, ωστόσο στην έκθεση, στη σελίδα 25 της εκθέσεως σας λέγεται ότι πλην των πιθανών συνεπειών δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες ε, συσχετισμός μάλλον μεταξύ τρορογμάτωσης και ε, δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν έχει τεκμηριωθεί. Αυτό λέτε. Επίσης επισημαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει σαν συνέπεια ε, πονοκέφαλο, αλλά εντάξει και εγώ παθαίνω πονοκέφαλο, αυτό σημαίνει πρέπει να εξορίσετε φυσικό αέριο, ίσως ελληνικό φυσικό αέριο. Καλώ λέει ο κύριο Λάνεν, όλε τι πτυχές βεβαίω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά εμεί είμαστε Επιτροπή περιβάλλοντο και πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα από την περιβαλλοντική σκοπιά. Η Ήτρε έχει κάνει σχετική ακρόαση, όπου ασφαλώ ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την ασφάλεια στην ε, προμήθεια ενέργεια, ε, τι ενεργειακές πτυχέ κτλ. Και αυτό καταλάβει στην έκθεσή τη. Εδώ την, έκθεση την έχουμε στήσει εμεί από τη δική μα την οπτική γωνία. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και παραξενεύομαι για την εξέλιξη, για την τροπή που έχει πάρει, τη λέει ο κύριο Έικχαουτ. Εμεί ω Επιτροπή Περιβάλλοντο πολύ συχνά ζητούμε ειδικέ εξειδικευμένε μελέτε για επιστημονικά θέματα, όπω έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση και έτσι ως ε, βουλευτές καλό θα ήταν τουλάχιστον, τουλάχιστον να ευχαριστούμε τους επιστήμονες που ήρθαν εδώ να μας προσφέρουν εκθεσή τους και να τους καταθέσουμε ερωτήσεις να έχουμε ερωτήσει, όχι να τους προσβάλλουμε και να επιτιθέμεθα στα όσα λένε. Γιατί αυτό δεν είναι τρόπος να φέρεται κανείς σε επιστήμονες και επιπλέον όταν γνωρίζει κανείς ότι στο Κορνέλ, το Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κέντρο Γιουτούμπελ έχουν επίσης καταλήξει μια πρόταση για μορατόριουμ και στο EPA επίσης υπάρχουν αμφιβολίες. Εάν λοιπόν όλες αυτές οι επιστημονικές μελέτες μελέτες καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα με την ε, έκθεση που συζητούμε, μήπως θα έπρεπε να διερωτηθούμε για το αν είναι κατάλληλο η επιλογή που έχουμε κάνει. Μην προσβάλλετε λοιπόν τον Αγγελία Φόρο. Ακούστε ποια είναι η επιστημονική βάση και μετά προχωρήστε στην πολιτική μετάφρασή της. Αυτό πρέπει να συστήσουμε εδώ. Πολιτική μετάφραση που μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που λέει η έκθεση. Αλλά αυτό συνεπάγεται μια πολιτική συζήτηση, μάλλον προϋποθέτει μια πολιτική συζήτηση. Εμείς ως πράσινοι λέμε ότι αποτελεί μια επιπλέον πέραν των υπολείπων απόδειξη η εν λόγω έκθεση ότι η λύση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου δεν είναι σωστός δρόμος. Αυτό. Πάντως ευχαριστώ πολύ τους επιστήμονες που μας δίνουν τις πληροφορίες. Τώρα, για να ξεφύγουμε από την επιστημονική συζήτηση, τώρα, ξεφύγουμε από την επιστημονική συζήτηση σημαίνει και να καταθέσουμε ένα ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στο κεφάλαιο 4, που κανεί δεν έχει ακόμη θίξει, βλέπουμε πολλά κενά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εντοπίζονται πολλά κενά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σκοπεύει να κάνει για το θέμα αυτό. Και εντωμεταξύ, τι σκοπεύει να αποφασίσει για, το, για τις προσπάθειες που αναπτύσσονται ανά την Ευρώπη για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί και αναγνωριστεί επισήμως και άρα θα πρέπει εμείς αντί να καταγγέλουμε για το λάθος μήνυμα τους ε, επιστήμονες, καλό θα είναι να ακούσουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Πολλές φορές ξέρουμε ότι οι επιστήμονε δίνουν μηνύματα που δεν μα αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε και να τα γνωρίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο Σταυρονικά. Κύριε Λουκοσέφσκα, έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων κυρίες και κύριοι, θα έλεγα ότι αυτή η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με την Ευρώπη σε τόσο υψηλό επίπεδο ότι καμιά χώρα δεν θα εισήγαγε κάτι επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον. Όμως μπορεί κανείς να συζητήσει με επιστήμονες, διότι αν δεν υπήρχαν αμφιβολίες, αν δεν υπήρχαν αναλύσεις με διαφορετικά αποτελέσματα δεν θα είχαμε συζήτηση και πολλές συζητήσεις αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες επιστημόνων με διαφορετικές απόψεις που διαφέρουν μεταξύ τους. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κάποιος ανέφερε και είπε εδώ ότι <clears throat> μια τοποθέτηση ενός, ε, μιας ομάδας λομπίστων υπέρ του σχιστολιθικού αερίου ε, προσέξτε, από τότε που ακούστηκε ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα συστολιθικού αερίου στην Πολωνία, υπάρχει και ομάδα που είναι και εναντίον. Είναι μεγάλη δουλειά, μεγάλο εγχείρημα αυτό, όπου κερδίζει κάποιος, κάποιοι άλλοι χάνουν. Και αυτό είναι ο λόγος ακριβώς πίσω από αυτήν την υπερβολική δραστηριοποίηση και δραστηριότητα. Ενώ υπάρχουν κάποιοι που είναι εναντίον, ενώ δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά κριτήρια που να λένε ότι είναι επικίνδυνη αυτή η δραστηριότητα. Και άλλοι είναι υπέρ, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια ελπίδα για το μέλλον να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας όσον αφορά την ε, χρήση φυσικών πόρων. Είμαστε κατά του ε, άνθρακα, κατά του, ε, της πυρηνικής ενέργειας, αν είμαστε κατά και του σχιστολιθικού αερίου, τότε υπέρ τίνος ε, υλικού ή στοιχείου είμαστε. Διαβάζουμε σε αυτή τη μελέτη και αναφέρεται στην αρχή-αρχή πιθανή επίπτωση, λέει, της υδραυλικής θράψης ή ρηγματοποίησης στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Και μετά ακούμε ότι υπάρχει τέτοια επίπτωση και επιρροή και στο περιβάλλον και στην υγεία. Ενώ στην μελέτη την ίδια δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ή αναφορά ότι κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει. Έχουμε την περίπτωση μιας γυναίκας που είχε ένα καρκίνο που παρουσίασε. Όμως η συνάρτηση αυτή, δηλαδή κάποιοι που ζουν κοντά σε ανεμόμυλους και αυτοί αρρωσταίνουν. Ε, τι θα συμφωνούσατε λοιπόν ότι εκείνοι που ζουν κοντά σε ανεμογεννήτριες ε, συναρτώνται αυτές οι περιπτώσεις ασθένειας και θα έπρεπε να απαγορεύθουν οι ανεμογεννήτριες που παράγουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την αιωλική δηλαδή ενέργεια ηλεκτρικό ρεύμα φυσικά όχι υπάρχει ανάγκη να διεξαχθούν συζητήσεις και διαβουλεύσεις χωρίς συναισθηματική φόρτιση και χωρίς προκαταλήψεις. Μια τέτοια μελέτη λοιπόν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ληφθεί υπόψη. Ο Κρήτον Αρσένης παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και για την Λίντα Μακάβεν και για το θέμα που συζητούν, πώς όλα αυτά εντάσσονται και πώς έγινε η κίνηση για αυτή τη νέα προοπτική του αερίου και του σχιστολιθικού αερίου. Πώς εντάσσεται αυτό και μπορεί να συνεργαστεί και να συνταχθεί με νέες πολιτικές χαμηλών εκπομπών ε, ρήπων διοξιδίου του άνθρακα σε ένα νέο ενεργειακό πλαίσιο. Και όπως ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι, υπάρχει, υπάρχουν κενά που μπορούμε να εντοπίσουμε. Και αυτή η μελέτη μας βοηθά να εντοπίσουμε κενά και ελλείψεις. Πρέπει να τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Πρώτον στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ακούγαμε επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται σε σχέση με την πρόταση αυτής της μελέτης. Ότι δηλαδή ακόμα και σε χώρες όπου παραδοσιακά υπάρχουν γεωτρήσεις που γίνονται για την αναζήτηση, τον εντοπισμό φυσικού αερίου και πετρελαίου, ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις και μήπως χρειάζεται μια οδηγία πλαίσιο για τέτοιου είδους δραστηριότητες, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν καλύπτουν την εξόριξη σε χαμηλότερο επίπεδο κάτω από 500.000 κυβικά μέτρα ημερήσια, μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι ως προς αυτά, αυτά τα πλαίσια και για την, ε, ε, το νερό και την οδηγία σε 2, για όλα αυτά τα χημικά και τις χημικές ουσίες που δεν καλύπτονται από αυτή την οδηγία και που σκοπεύουν να τις χρησιμοποιήσουν λέει αυτές οι εταιρείες χωρίς να είναι και γνωστή κιόλα η χρήση τους ή να γνωστοποιείται και για την οδηγία πλαίσιο για το πώς πρέπει να επανεκτιμηθεί και να αξιολωθεί όσον αφορά το νερό για τέτοιου είδους γεωτρήσεις ε, όσον αφορά την, ε, τον θρηματισμό και τον, ε, την ρηγματοποίηση. Θα ήθελα να ακούσουμε τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολλά τα στοιχεία για να προβληματιστούμε και να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάθος, σε λεπτομέρειες και να τα ξανακοιτάξουμε την οδηγία για παράδειγμα πλαίσιο για το νερό, για τους υδάτινους πόρους. Να τα ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, βρισκόμαστε τώρα στην λήξη του χρόνου, πολύ κοντά στην λήξη του χρόνου. Έχουμε άλλους έξι που έχουν εγγραφεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να παρέμουν, λυπούμε. Είναι όμως δίκαιο να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Άλτμαν. Η Επιτροπή δεν ήθελε σήμερα να τοποθετηθεί. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες όπου θα μπορεί να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσατε τις ερωτήσεις που υπάρχουν κύριε Άλτμαν. Θα θέλατε τώρα να λάβετε τον λόγο για να απαντήσετε σύντομα για αυτές τις τοποθετήσεις που έγιναν κατά της μελέτης σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ασφαλώς είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Ενδιαφέρον θέμα. Και από καθαρά η επιστημονική απόψη ήταν ενδιαφέρον ότι αναλάβαμε μας με τους συναδέλφους να εκπονήσουμε τη μελέτη. Υπήρξαν ερωτήματα ως προς την ανεξαρτησία της επιχείρησης την οποία, στην οποία Η εταιρεία μας συντηρήθηκε το 1982 πρέπει να σας πω. Έχουμε περίπου 30 χρόνια εμπειρία. Ο στόχος δε, κατά την ε, ίδρυση της εταιρεία ήταν ε, να ε, εστιαστούμε κυρίως σε θέματα αηφορίας, γεωργίας, κινητικότητας. Εντάξει, η λέξη αηφορία δεν υπήρχε τότε ακόμη, αλλά αυτό ήταν ο στόχος μας και αυτό και πράξαμε. Εργαστήκαμε και πάνω σε θέματα συμβατικών μορφών ενέργειας, φυσικό αέριο, Φερρυπίν. Άνθρακα και άλλες πηγές. Νομίζω ότι μπορούμε δηλαδή να ισχυριστούμε πως είμαστε ανεξάρτητοι. Κάτι άλλο επίσης. Αναφέρθηκε πως έχουμε εμπορικό συμφέρον, έχουμε οικονομικό συμφέρον από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουμε κανένα κέρδο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εργαζόμαστε ω ανεξάρτητοι επιστήμονες και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να τις ε, διαβάσει. Αυτό ε, συμπεριλαμβάνει και πετρελαϊκές εταιρείε και αυτοκινητοβιομηχανία και επιχειρήσεις που ασχολούνται με το φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο. μπορείς να μην γνωρίζετε τα ονόματα όλων των πελατών μας, πάντως είναι όλοι μεγάλοι γνωστοί διεθνείς επιχειρήσεις δηλαδή. Έχουμε εργαστεί με πολλούς ε, πελάτες όπως και θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ε, ε, διοικήσεις και ως εκ τούτου δεν αμφισβητείται νομίζω, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ουδετερότητά μας. Και ίσως κάνετε τον κόπο να δείξετε μια ματιά στο έγγραφο αυτό είναι τιμή για μένα το ότι κάποιος κάθισε να διαβάσει και να αναλύσει με τόσο μεγάλη προσοχή τα 20 άτομα που απαρτίζουν την επιχειρήση μου. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε εμπορικό χαρακτήρα, δεν κερδίζουμε δηλαδή από αυτά που λέμε. Σε σχέση με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και την, ε, την αγοραία αξία από τη Γερμανία σε σχέση με την Gazprom. Κοιτάξτε, εμεί δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε καμία οικονομική αξιολόγηση, οικονόμηση επιχειρησιακών ευκαιριών και τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν το έχουμε πράξει αυτό. Παρακαλώ λοιπόν μην θεωρείτε ότι υπάρχει οικονομική ανάλυση στην έκθεσή μας. Εμείς ούτε διανοηθήκαμε να κάνουμε ανάλυση του κατά πόσον από ε, άποψη οικονομική ή επιχειρηματική θα ήταν σκόπιμο στην Ευρώπη, θα είχε δηλαδή θα ήταν συμφέρον στην Ευρώπη να γίνει εξόριξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Ε, αυτό πρέπει να είναι σε Και επίσης ε, για τις άλλες πτυχές που συστήθηκαν εδώ, που ακούστηκαν, είμαι στη θέσή σας για κάθε συζήτηση επί της ουσίας ε, για τα δεδομένα, για τα συμπεράσματα, για τη βάση πάνω στην οποία κάνουμε την ανάλυση μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η πολύ σημαντική συζήτηση καθήκον τη επιτροπή μας άλλωστε ήταν να τη ξεγάγουμε και θα δούμε πώ θα χειριστούμε το θέμα περαιτέρω. Ο κύριο Σόνικ μου λέει ότι αυτό το έγγραφο των Πολωνών επιστημόνων θα σα διατεθεί, θα δώσει και το όνομα το οποίο χρήσιμο να σας καταγράψει η γραμματεία. Θα ενημερωθούμε 17-18 είναι θέματα που θα δούμε αύριο προς το τέλος της συνεδρίας που μάλλον θα έχουμε αρκετό χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και θα κλείσουμε προς το παρόν τη συνεδρία. Χαίρετε. Okay. Thank you.